προδιαγραφ... τις διατάξεις του άρθρου 7 της ε, Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και τέλος, ε, προτάθηκε μια συμβιβαστική λύση όσον αφορά τις ε, εκτελεστικές πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε να ακολουθηθεί το άρθρο 6 παράγραφος 4 όμως για το θέμα αυτό χρειάζεται μία έκτακτη συνεδρίαση και τα τρία θεσμικά όργανα κατάφεραν να συμφωνήσουν σε μια συμβιβαστική λύση όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία ελέγχου για την εφαρμογή του κανονισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, καθώς επίσης και για την διαδικασία ελέγχου διασφάλισης, ότι δεν θα ανταλλάσσονται δεδομένα ανάμεσα στο σύστημα e-call και σε άλλες παρόμοιες υπηρεσίες διότι γι' αυτό προβλέπονται οι εκτελεστικές πράξεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητέ τη Επιτροπή ΕΛΥΜΠΕ, καθώς και όσους συμμετείχαν στον τριμερή διάλογο, ιδιαίτερα την ε, Γραμματεία, η οποία βοήθησε και στήριξε πάρα πολύ το έργο μα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Άξελ. Επόμενο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να ενημερωθούμε είναι για την Europol. Έγινε ε, στις 8 Δεκεμβρίου τριμερής διάλογος και ο κύριος Δία Δεμέρα δεν μπορεί, ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα και μου ζητάει να σας ενημερώσω. Κατά τον τριμερή διάλογο συζητήθηκαν ε, τα εξή ζητήματα, διαδικασία για το διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και οι διατάξει για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τα δύο ζητήματα είναι στον πυρήνα αυτού του φακέλου. Πώς ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορεί να ελέγχει το έργο αυτού του σημαντικού οργανισμού. Είναι θέμα δημοκρατίας, πρέπει να είναι κάποιος υπόλογος και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο μας. Ε, και για τα δύο ζητήματα ακόμη δεν είναι ορατός ο κάποιος πιθανός ε, συμβιβασμός στα τρία θεσμικά όργανα. Πάντως ο εισηγητής ε, και ο σκιώδης είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για αυτό τον κανονισμό της Europol θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες διατάξεις σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον έλεγχο του έργου της Europol. Το, στις αρχές Φεβρουαρίου, στον επόμενο τριμερή διάλογο, έχει προβλεφθεί η σύσκεψη για τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων για την κανονισμό της Europol. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η ενημέρωση. Ας περάσουμε στη ψηφοφορία τώρα. Χρειάζεστε την κάρτα ψηφοφορίας. Ελπίζω να την έχετε όλοι μαζί σας. Η κατάσταση στην Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση. Στις 5 Νοεμβρίου στη Λίμπη, όπως ξέρετε, ψηφίσαμε την προφορική ερώτηση που μας οδηγεί σε αυτή την ψηφοφορία. Η συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έγινε τον Νοέμβρη στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνατε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μία είναι η ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία, πέρας. 37 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν σκληρά. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο. Οργανισμός ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση για την επιβολή του νόμου. Σε πόλ θα ζητήσω από τον συνάδελφο Γιάννα Άλμπρεχτ. Εγώ δυστυχώς θα πρέπει να... Ε, να... Να φύγω κάποια στιγμή. Θα ζητήσω λοιπόν από τον συνάδελφο να προεδρεύσει. Dear colleagues, we start with... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε με το σημείο 7, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, ΣΕΠΟΛ. Η συγγήτριά μας είναι η Κίνγκα Γκάλ. Και εδώ θα συζητήσουμε το, το σχέδιο έκθεσης και την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών, η οποία είναι η 8η Ιανουαρίου. Στις 5 Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα της ΕΣΕΠΟΛ στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Δεν είναι ένα, μια, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με την παραδοσιακή έννοια. Ή αφορά την ε, πανευρωπαϊκή συνεργασία και κατάρτιση αστυνομικών. Υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια κατάρτιση, διότι πολλοί αξιωματική επιβολή του νόμου χρειάζονται κατάρτιση για, τα νέα, για τις νέες μεθόδους. Η κατάρτιση αυτή επίσης μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην πολιτική θεωρία, στην θεωρία και την πράξη. Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία που μπορεί να επιφέρει σε πόλη είναι η μεγιστοποίηση ε, της ε, σχέσεις κόστους όφελους και ο ίσως καταμερισμός της εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι που χρειάζεται. Ο ισχύων κανονισμός εξυγχρονίζει τη νομική βάση της ΕΠΟΛ, κάτι που χρειαζόταν ε, μετά από τις αλλαγές που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία έδωσε στην ΣΕΠΟΛ νέες αρμοδιότητες και το Κοινοβούλιο ζήτησε αρκετές φορές την τροποποίηση και τον εξυγχρονισμό του κανονισμού αυτού. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καλωσορίσω αυτήν την νέα ε, πρόταση, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στη ΣΕΠΟΛ να εφαρμόσει αποτελεσματικά το νέο ε, σχέδιο κατάρτισης των Ευρωπαίων αστυνομικών. επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό η δομή, κύρια δομή τη ΕΠΟΛ να παραμείνει ω έχει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει μια πολύ ισχυρή θέση για την διατήρηση της ΣΕΠΟΛ ε, και του καθεστώτος της ΕΠΟΛ και στηρίζουμε την προσπάθεια και τη συνεισφορά της ΕΣΕΠΟΛ για την δημιουργία μιας πραγματικής ε, κουλτούρας επιβολής ε, του νόμου στην Ευρώπη. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσει η ΕΣΕΠΟΛ στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να εστιάσει τους περιορισμένους πόρους της σε συγκεκριμένα ε, σημεία που θα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο συντονιστικός και υποστηρικτικός ρόλος της ΕΠΟΛ. Οι τροπολογίες λοιπόν που κατέθεσα είναι σχετικές με αυτά και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω πολύ τη Γραμματεία για τη βοήθειά της. Για να διασφαλιστεί λοιπόν η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπο τη ΕΠΟΛ, οι περιορισμένοι πόροι τη θα πρέπει να εστιάσουν σε συγκεκριμένου τομεί με συγκεκριμένη και ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ακόμα περισσότερε αρμοδιότητε. Χρειάζεται αποτελεσματικότερος συντονισμός ανάμεσα στις ε, υπηρεσίες έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σωστά και αποτελεσματικά οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, να εκμεταλλευτούμε τις ε, συνέργειες και να αποφύγουμε την διπλή δουλειά όπου μπορούμε. Επίσης, η πόλη θα πρέπει να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την ε, βοήθεια και την υποστήριξη του έργου της αστυνομικής συνεργασίας και πιστεύω ότι χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση για την ΣΕΠΟΛ και πιστεύω επίσης πως ο προτινόμενος προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στο έργο και τις νέες αρμοδιότητες της ΕΠΟΛ. Χρειάζεται λοιπόν αύξηση του προϋπολογισμού και όπως είπα, συντονισμός και καλύτερη εφαρμογή της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και ξεκάθαρη εντολή της ΕΣΕΠΟΛ και υπάρχουν οι αντίστοιχες τροπολογίες που κατέθεσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία της υπηρεσίας αυτής και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η ΣΕΠΟΛ θα πρέπει να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να ενισχύσει τον συντονισμό και όχι μόνο να ασκεί υποστηρικτικό έργο. Και υπάρχουν επίσης και οι αντίστοιχες τροπολογίες για τα θέματα αυτά. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι οι περιορισμένοι πόροι της ΕΠΟΛ θα πρέπει να εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς που θα έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και θα έχουν διασυνοριακή διάσταση. Αυτές είναι οι τροπολογίες εν ολίγης. Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με τους κοιόδης συζητητές και να συζητήσω με εκείνους και με όλους τους ενδιαφέρομενους. Σας ευχαριστώ. Uh, ευχαριστούμε κυρία Γκάλ. Τώρα μόνο ένας συνάδελφος, μία συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο, κυρία Βίξτρομ. Αν κάποιος άλλο θέλει να συμμετάσχει, παρακαλώ να μου το πείτε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ε, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες αναφορές στις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή προοπτική. Συμφωνούμε απολύτως εδώ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να καλύπτονται από όλε τι δραστηριότητε τη ΣΕΠΟΛ. Γι' αυτό η τροπολογία 7 της εισηγήτριας είναι πρόσδεκτη είναι σημαντικό να το καταλάβει βέβαια αυτό και η ΣΕΠΟΛ, γιατί ω τώρα έχουμε ακούσει διαφορετικά πράγματα από την Ακαδημία. Ευτυχώ λοιπόν που το διευκρινίζει η συγκήτρια. Οι δραστηριότητε τη ΣΕΠΟΛ θα πρέπει να επικεντρώνονται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να μην υπάρχει επικάλυψη με την εθνική εκπαίδευση. Επίση, είναι σημαντικό και συμφωνώ πολύ με την εισηγήτρια ότι όταν αναθέτουμε νέε αρμοδιότητε στην Ακαδημία θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει και η ανάλογη χρηματοδότηση. Σημαντικό είναι τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Είμαι και πάλι υπέρ της συγχώνευσης της ΕΠΟΛ με την Europol ή τουλάχιστον να βρίσκονται στην ίδια έδρα ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία τους και να υπάρξει οικονόμηση χρημάτων. Παροτρύνω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει μια και καλή ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος ε, ε, του ορισμού της έδρας της Apple στην Βουδαπέστη αντί να ε, μείνει μαζί με την Europol στη Χάγη. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω την συγκεκριμένη γιατί θέλει στο άρθρο 3 να διαγραφούν οι τροπολογίες 8 και 9. Θα ήταν καλό η εκπαίδευση που παρέχει η Apple να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερους αστυνομικούς με, με κοινό εκπαιδευτικό τίτλο, ε, κύκλο. Συγγνώμη και εκπαίδευση. Επίσης, λίγη σύγχυση μου προκαλεί η τροπολογία 12 με την κοινή επιστημονική έρευνα, που, όπου η συγγήτρια άλλαξε το «σαλ» πρόκειται σε ένα πολύ πιο αδύναμο μέι. «δύναται». Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να μείνει ο όρος «σαλ», «δύναται». Μάλλον ναι, πρόκειται. Επίσης ό,τι αφορά τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Ακαδημίας, πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης να ξεκινήσουμε αντιμετωπίζοντα τα πράγματα από την πλευρά των αναγκών και να υπάρχει ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα τη δικαιοσύνη και τη αστυνομική συνεργασία. Βεβαίω, προφανώ. Πάνω απ' όλα σε συμφωνία με τι κοινέ μα αξίε. Θα έπρεπε δηλαδή να δούμε πώ χρειάζεται περισσότερη ευθυγράμμιση με τα θεμελιώδη ανθρωπίνα δικαιώματα, του στόχου και τι αρμοδιότητε τη Ακαδημία στις διατάξεις για την εκπαίδευση από την οδηγία ε, για τα δικαιώματα των θυμάτων. Και αυτό πρέπει να το επεξεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κατάλογό μας, οπότε θα ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ έχω ουσιαστικά κάτι να προσθέσω σε σχέση με την παρουσίαση που έγινε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, την, ε, το περασμένο μήνα. Ε, σημείωσα λοιπόν τα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε πάλι την εισηγήτρια και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σεσίλια για την συνεργασία. Οι τροπολογίες 8 και 9 έχουν ως στόχο να είναι αποτελεσματική η αστυνομική ακαδημία διότι είναι περιορισμένοι οι πόροι και άρα θα πρέπει να επικεντρωθούν σε κάποιους θεματικούς τομείς που παρουσιάζουν μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ποιότητα και ελκυστικότητα. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Τροπολογία 9. Τροπολογία 12 τώρα. Μπορούμε να το συζητήσουμε το ΣΑΛ και το ΜΕΙ. Δεν έχω πρόβλημα να μετατρέψουμε την δυνητική διάταξη σε ε, καταφατική με το ΣΑΛ. Ε, για το θέμα του τρόπου έχει κλείσει η συζήτηση, ε, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έδρα, αν θέλετε. Ε, ευχαριστώ πάντως για την καλή συνεργασία που είχαμε. Η κυρία Βίξτρομ, για δεν καταλαβαίνω να μας δίνει τέτοια απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού της έκανε συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω νούμερα. Θέλω να ξέρω ποιο είναι το κόστος, ποιες επιπτώσεις υπάρχουν από οικονομικής πλευράς για τον οργανισμό. Αγενής είναι, όχι μόνο ε, άσχετη με το θέμα. Εγώ κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση και τι ε, ε, με πλήρη διαφάνεια θα μας δώσει κάποια στιγμή απάντηση. Λίγο περίεργα δεν είναι όλα αυτά. Έχει τίποτα να πει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Φυσικά με απόλυτη διαφάνεια θα απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Φυσικά, καταγράψαμε το ότι ενδεχομένω ο συνομοθέτη θα καταθέσει νέα πρόταση και φυσικά σημειώσαμε ε, το έτοιμά σα για την εκτίμηση του κόστου για τη μεταφορά της έδρα στη Βουδαπέστη. Φυσικά θα σα απαντήσουμε. Περασμένη φορά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ε, είχαμε ήδη σημειώσει το ίδιο ερώτημα. Ζητώ συγγνώμη που εκλαμβάνεται ως εγενής η προηγούμενη απάντησή μου δεν ήταν η πρόθεση μου. Μόνικα Χολμαϊ. Μπορώ να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ε, η επιλογή της Ουγγαρίας έγινε διότι η Ουγγαρία ήδη δήλωσε μία προθυμία να αναλάβει το ε, μεγαλύτερο μέρος του κόστου του για το ενίκιο για τη στέγαση της αστυνομικής ε, ακαδημίας. Κάτι που δεν έδειξε η κυβέρνηση των 100 χωρών η οποία δεν ήθελε να αναλάβει κανένα κόστος. Γι' αυτό λοιπόν έγινε η επιλογή Τη ε, Βουδαπέστη, της Ουγγαρίας, διότι το κόστος ήταν πάρα πολύ χαμηλότερο από εκείνο που θα υπήρχε αν η ΣΕΠΟΛ πήγαινε στη Χάγη. Γι' αυτό λοιπόν έγιναν αυτά και φυσικά πρέπει να διασφαλιστεί καταρχάς τη ασφάλεια της ε, ΣΕΠΟΛ, η ασφάλεια των εκτηρίων, τα οποία ήταν ήδη διαθέσιμα. Για την ε, μετακόμιση της ΕΠΟΛ στη Χάγη θα χρειαζόταν ένα επιπλέον κτίριο και αυτό θα επέφερε και επιπλέον κόστος. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε από το Συμβούλιο να πάει σε πόλη στην Ουγγαρία και μετά από 10 χρόνια θα επαναξεταστεί το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα παρόλα αυτά υποβάλλουμε και πάλι το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτό το χρόνο θα απαντηθεί. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση. Και να ξέρετε ότι για τις τροπολογίες η 8 Ιανουαρίου στις 12 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστούμε. Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο. Στις 27 Νοεμβρίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόταση για οδηγία για την προσωρινή νομική αρρωγή για υπόπτους ή κατα... κατηγορουμένους ε, με ποινή στέρησης ελευθερίας βάσει το άρθρο 82.2β της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής είναι ένα δεύτερο πακέτο για διαδικαστικά δικαιώματα, ώστε να ολοκληρωθεί ο δικός χάρτης για την ενίσχυση των ε, διαδικαστικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων σε ποινικέ διαδικασίες. Στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία υπήρξε ένα έγγραφο εργασία από τον εισηγητή μα κύριο Ντιγιάνγκ το Μάρτιο δηλαδή του 2014 για να ξεκινήσει η συζήτηση στη ΛΥΠΕ έχει αρχίσει τι εργασίε στο Συμβούλιο, αλλά δεν έχει ακόμα εγκρίνει μια γενική προσέγγιση. Ο κ. Ντένι Δεγιόν επαναδιορίστηκε συγγνώμη, εισηγητή για την 8η κοινοβουλευτική θητεία. Στι 11 Νοεμβρίου θα ήθελα να σα θυμίσω θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για αυτή την πρόταση και για τι άλλε προτινόμενε οδηγίε για το τεκμήριο αθωότητα και για τα παιδιά ε, υπόπτωση και κατηγορουμένους ε, στις ποινικές διαδικασίες. Θα παρουσιάσει ο κ. Ντεγιόν τώρα το σχέδιο έκθεσης. Αν είστε έτοιμος, παρακαλούμε. Ντένις. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Με συγχωρείς κιόλας που καθυστέρησα λιγάκι γιατί είχα κάποιες συζητήσεις. Δεν θα σας πω γιατί. Δεν έχει σημασία η έκθεση για την νομική αρρωγή. Λοιπόν, ε, πιστεύω πως αξίζει ένα, μια ιστορική αναδρομή για το πώς κατέληξα σε αυτήν την έκθεση και πιστεύω πως είναι καλύτερο αυτό παρά να σας αναφέρω τις ε, επιμέρους τροπολογίες. Αν ε, συζητήσετε με τα διάφορα Υπουργεία Δικαιοσύνη στην Ευρώπη ή με τις αρχές επιβολής του νόμου θα δείτε ότι πάρα πολλοί έχουν ε, δηλώσει την ευχαρίστησή τους για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης γιατί επιφέρει πολύ γρήγορα αποτελέσματα και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Ωστόσο, η όλη προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι ότι οι αρχές επιβολής του νόμου για να έχουν λοιπόν αυτά τα επιθυμητά περισσότερα αποτελέσματα στον τομέα της συνεργασίας δεν ακολούθησαν αυτόν τον κατάλογο των δικονομικών δικαιωμάτων και υπάρχει ο δικός χάρτης για τα δικονομικά δικαιώματα. Όμως η διαδικασία του οδικού αυτού χάρτη είναι χρονοβόρος. Έχει πολλά στάδια και έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου δεν έχουν ακολουθηθεί αυτά τα στάδια. Άτομα στα οποία δεν χορηγήθηκε δικηγόρος, δεν χορηγήθηκε διερμηνία, δεν μιλούσαν τη γλώσσα και προσπαθούμε λοιπόν να συμπληρώσουμε τις ελλείψεις και στο μεταξύ δεν υπάρχει καμία ε, εγγύηση για την ε, διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων σε όσους ε, συλλαμβάνονται με το Ευρωπαϊκό Ανταλμά Σύλληψης. Η προσέγγιση που είχαν ακολουθήσει όλα τα θεσμικά όργανα ε, ήταν μια προσέγγιση με την οποία κανείς δεν έμεινε ευχαριστημένος και ιδιαίτερα όχι το Κοινοβούλιο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια διτή προσέγγιση. Από τη μία προσπαθούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία για να ε, διασφαλιστούν και τα δικονομικά δικαιώματα των κατηγορουμένων υπόπτων και εξητούμενων και από την άλλη, την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είδαμε και εξετάσαμε με ε, λεπτομερώς το πώς λειτουργεί αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και πώς μπορούμε να εισαγάγουμε περισσότερες ε, ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν έχουν δοθεί τέτοιε ασφαλιστικές δικλείδες προς το παρόν, αλλά ελπίζουμε να γίνουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται περισσότερη πίεση για τις δικονομικές ασφαλιστικές δικλείδες και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα και με τρόπο ολοκληρωμένο και όχι κατακαιρματισμένο. Και με βάση όλα αυτά, συνέταξα την έκθεσή μου διότι δεν μου ευχαριστεί καθόλου αυτή η κατακαιρματισμένη προσέγγιση του οδικού χάρτη. Όμως, στο θέμα της νομικής αρρωγής, μία οδηγία και μία σύσταση θα κατακαιρματίσει ακόμα περισσότερο την ε, κατάσταση. Χρειάζεται κάτι πολιτικά, χρειάζονται πολιτικές εδεσμεύσεις, διότι χωρίς αυτές το πρόβλημα εντείνεται και αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε για τα δικονομικά δικαιώματα βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν έχει τις διασφαλίσεις που θα έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε τουλάχιστον να διασφαλίσουμε την ύπαρξη των ε, αναγκαίων, δηλαδή το δικαίωμα νομικής αρρωγής στα πρόσωπα, στην ε, οδηγία, να αναφερθούμε τουλάχιστον, αν όχι να διευκρινίσουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας νομικής αρρωγής και χρειάζεται η διασφάλιση. Θα μπορούσαμε ίσως να το κάνουμε αυτό με μία αναφορά στην ανάγκη περισσότερων δικονομικών δικαιωμάτων. Γενικά δεν συμφωνώ καθόλου όπως βλέπετε με αυτόν τον κατακαιρματισμό και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει οδηγία πρόσβαση σε δικηγόρο και εφόσον αναγνωριστεί το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, η νομική αρρωγή δεν ε, μπορεί να είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτό. Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή που διέπει αυτό αυτές ε, τις τροπολογίες. Λοιπόν, λιγότερος κατακαιρματισμός και εφόσον αναγνωρίσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο δεν μπορούμε να ε, λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν το, τη δυνατότητα ε, να πληρώσουν δικηγόρο δεν θα έχουν και δικαίωμα πρόσβαση σε αυτόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζει το δικαίωμα αυτό και γι' αυτό στη δική μου έκθεση προσπαθώ να το αντιμετωπίσω και γι' αυτό αναφέρω ότι χρειάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο κατακαιρματισμό και υιοθετώ αυτή την προσέγγιση. Ότι αν δηλαδή έχει το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, πρέπει να έχει το δικαίωμα και σε νομική ερωγή. Φυσικά σέβομαι απόλυτα τις διαφορές των κρατών μελών στο ζήτημα τη νομική αρρωγή. Και πρέπει να διασφαλιστεί ένας ε, δικηγόρος μιας ε, κάποιας ποιότητας και όχι κάποιος ασκούμενος ο οποίος ε, δεν πληρώνεται. Υπάρχει λοιπόν αρκετό πεδίο ελιγμών για τα κράτη-μέλη, διότι όπως είπα σέβομαι τις διαφορές των νομικών συστημάτων, όμως υπάρχουν οι αντίστοιχες οδηγίες και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και για την ποιότητα του ε, συνηγόρου. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να παρουσιάσω ένα δίκαιο πακέτο. Γνωρίζω βέβαια πως ε, δεν κινούνται και πολύ γρήγορα τα πράγματα στο Συμβούλιο, ελπίζω όμως αυτό να αλλάξει τους προσεχείς μήνες. Και επίσης ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη, όμως δεν μπορείς να έχεις την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Εάν θέλεις ένα ολοκληρωμένο έταλμα σύλληψης πρέπει να ε, διασφαλίζεις και την πλήρη γάμα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και να αναγνωρίσεις επομένως το δικαίωμα στη νομική αρρωγή. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και με την έκθεσή μου. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις αντιδράσεις σας και να σας πω ότι δεν πρόλαβα να διοργανώσω συνάντηση των σκιωδών εισηγητών ακόμα αλλά πιστεύω πως με το που θα γνωρίζουμε τη θέση του καθενός θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεδριάσουμε, να συναντηθούμε πολλές φορές, να τα συζητήσουμε διεξοδικώς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ζητούν το λόγο η κυρία Σίπελ, η κυρία Σαρχεντίνη. Παρακαλώ να σκούνται τα χέρια σας. Ο λόγος στην κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ντένις αναφέρθηκε σε πάρα πολλά σημεία, γι' αυτό και εγώ θα περιοριστώ σε ορισμένα από αυτά. Η εντύπωση που αποκόμισα από αυτό το διπλό πακέτο δικονομικών δικαιωμάτων είναι ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ίδιες πολύ περιορισμένες και αυτό ισχύει και για τις ε, τρεις ε, διαδικασίες. Εάν θέλουμε μια διαφορετική διαδικασία για ορισμένες ομάδες όπως τα παιδιά για παράδειγμα πρέπει να ε, αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ε, νομική αρρωγή. Πρέπει να επεκταθεί πολύ περισσότερο και αυτό ισχύει και για το δικαίωμα σε δικηγόρο. Πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τένις για την πολύ καλή δουλειά του. Παρότι δεν έχουμε προλάβει να συναντηθούμε οι σκιώδεις εισηγητές, υπήρξε κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο μία ανταλλαγή απόψεων αρκετά περιεκτική. Πιστεύω σε γενικές γραμμές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε μεν στην νομική αρρωγή, αλλά και στο δικαίωμα ε, στη νομική αρρωγή. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω πως θα έπρεπε να ε, αναφέρεται στην οδηγία και όχι σε μία απλή σύσταση λόγω των διαφορών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική η νομική αρρωγή χρειάζεται να αναφερθούν και αυτές και επίσης να γίνουν σεβαστές και οι επιθυμίες ε, για την επιλογή έμπιστου δικηγόρου στα πλαίσια της νομικής αρρωγής. Πρέπει να δοθεί επίσης μια τέτοια διασφάλιση και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ναι μεν υπάρχουν διαφορές στα νομικά συστήματα των κρατών μελών όμως υπάρχει και η ανάγκη από τη στιγμή που κάποιος είναι κατηγορούμενος να έχει το δικαίωμα νομικής αργής και όχι αργότερα. Πρέπει η βοήθεια να είναι διαθέσιμη τη στιγμή που ο κατηγορούμενος ύποπτος τη χρειάζεται. Επίσης, η δυνατότητα και μόνο μίας αποζημίωσης του κόστους του δικηγόρου είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να φροντίσουμε να ε, μην ζητούνται αποζημιώσεις εκ των υστέρων. Είμαι σίγουρη πως σίγουρα θα καταθέσω και εγώ και άλλοι τροπολογίες για επιμέρους λεπτομέρειες, όμως πραγματικά περιμένω μια πολύ επικοδομητική συνεργασία με όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές, έτσι ώστε μαζί να ε, διατυπώσουμε και να υιοθετήσουμε μια πολύ ισχυρή στάση απέναντι στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν είχα δει την κυρία Μετσόλα μας. Έχει εξαρχίζει τη το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ρασίδα δεν μπορούσε να έρθει, γι' αυτό θα παρουσιάσω τη θέση της, είναι θέση της ομάδας μας για αυτή την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ντένις Δε Γιάνγκ για την δουλειά που έκανε για το σχέδιο έκθεσης. Με προσοχή διάβασα τις τροπολογίες του. Προς το παρόν δεν έχει συγκαλέσει σύσκεψη για τους κοιόδης. Προσβλέπω στη συζήτηση με τους υπόλοιπους κοιόδης. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή και πιστεύω ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Όμως προσοχή στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να είναι ισοσκελισμένη η πρόταση για το πεδίο εφαρμογής. διευρύνεται ε, το πεδίο ε, για την παροχή νομικής ε, αρρωγής σε όλους και όχι μόνο εκείνους στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, σε όλους τους υπόπτους και σε όλους τους κατηγορουμένους. Θέλουμε να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα για τα δικονομικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι τη νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου για τους συμπολίτες μας. Θέλουμε να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν ε, έχουμε όμως την αρμοδιότητα να θεσπίσουμε ένα σύστημα αυστηρό που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Είμαστε ρεαλιστές. Δεν θα πρέπει να παραβιάσουμε την κυριαρχία των κρατών μελών. Ας ακολουθήσουμε μόνο τη δική μας αποστολή, μην εμπλακούμε σε, περιτούς, ε, σε περιττές μάχες με το Συμβούλιο, εάν τα θέματα δεν άπτωται τις δικής μας αρμοδιότητες. Θέλετε και σε να εξασφαλίσετε την ποιότητα στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Συμφωνώ. Όμως, αναλογικότητα. Πρέπει να είναι αναλογικά αυτά που θα προτείνουμε κατόπιν. Θέλετε να διαγράψετε την ε, αναφορά στα δεδομένα Ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν έχει ασκηθεί αυτό το δικαίωμα για νομική αρρωγή, εγώ θέλω να παραμείνει αυτή η αναφορά. Είναι κέρια σημασία ώστε να είναι σε θέση τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος παροχής νομικής αρρωγής. Στη συνέχεια υπάρχει ειδική μνήμα για τα δικαιώματα των παιδιών για νομική αρρωγή και έχετε τελικά διαγράψει στο τελευταίο σχέδιο την ε, διάταξη αυτή. Μπορείτε να εξηγήσετε για ποιο λόγο. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τρίτον, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την παροχή νομικής αρρωγής θα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικότερα, λεπτομερέστερα. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος αυτός ο στόχος. Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με τον κύριο Ντε και τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές ούτω ώστε να είναι συνενετική και κρατεία η θέση στην οποία θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ. Σαρτζεντίνη, πράσινη. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Τένις Δεγιό για την ενδελεχή παρουσίαση του ζητήματος. Εκτιμώ το ότι έχει ως στόχο να παρέχεται η νομική αρρωγή από την αρχή της διαδικασίας και το ότι θέλει να επεκτείνει ε, το πεδίο εφαρμογής ε, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Νομίζω ότι είναι σωστό να αναλάβει την πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντισταθμίσει την αδράνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουμε πρόσβαση σε το εργαλείο. Ε, είμαστε και οι δύο Ολλανδοί και μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μα και γνωρίζουμε τι σημαίνει ε, νομική αρρώγη. Μπορεί κανεί στην αρχή να έχει δικηγόρο, συνήγορο, αλλά άμα ολοκληρωθεί η δίκη πρωτοβαθμίως, ε, δεν υπάρχει πλέον ε, νομική αρρωγή. Πρέπει να ξεκινήσει κανείς από την αρχή στο δικαστήριο δεύτερου βαθμού. Επίσης, ρωτήθηκε αν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στο τέλος της διαδικασίας. Πρέπει να δούμε, όπως είπε η κυρία Ζήπελ, τι ε, θα κάνουμε και αν θα δώσουμε την εντύπωση ότι αν κανείς δεν έχει χρήματα στο τέλος μιας δίκης, Ε, θα πρέπει παρόλα αυτά να ε, υποχρεωθεί να επιστρέψει χρήματα. Δεν θα μπορεί να ξεκινήσει καν την προσφυγή του γιατί θα ξέρει ότι δεν έχει χρήματα στο τέλος για να την καλύψει. Έπειτα για την νομική αρρωγή σε παιδιά. Νομίζω ότι στην οδηγία για τα παιδιά, την παιδική ηλικία που ήδη έχουμε συζητήσει, η νομική αρρωγή είναι θέμα εθνική αρμοδιότητα. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βέβαια πλέον λογική λύση, διότι πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να οργανωθεί έτσι η νομική αρρωγή που να μην ε, υπόκειται, να μην εξαρτάται από το φορέα κράτος. Επίσης, πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, η, η οδηγία για τα παιδιά και την νομική αρρωγή πρέπει να ε, ενδεχομένω να συνδυαστούν για να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα που να λειτουργεί εύρυθμα. Εγώ φοβάμαι ότι αν ορίσουμε πολύ χαμηλά τα όρια για τι ελάχιστε απαιτήσει μα, όπω το δικαίωμα σε συνήγορο, θα είναι πολύ ωραία στα χαρτιά όλα αυτά, όμω στην πράξη δεν θα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Διότι δεν θα υπάρχουν τόσοι δικηγόροι ελεύθεροι ή οι αμοιβέ θα είναι τόσο χαμηλέ για του δικηγόρου που κανεί δεν θα θέλει να αναλάβει. Θα γίνει δηλαδή κάτι σαν φιλόπτωχο το όλο σύστημα. Ο μόνο τρόπο για να προχωρήσουμε είναι να έχουμε μια σειρά από, έργο, ε, από συγκεκριμένα νομικά εργαλεία. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα δικηγορικό γραφείο και μια σειρά από υποθέσεις όπου θα μπορούν να παράσχουν αρρωγή. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί δικηγόροι στην Ολλανδία που δεν δέχονται να παράσχουν νομική αρρωγή, διότι είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβέ τους. Και έπειτα η άλλη λύση δεν είναι να στέλνουμε τους φοιτητές νομικής ε, για την ε, νομική αρρωγή γιατί κοστίζουν λίγο, διότι αυτό σημαίνει διακριτική μεταχείριση. Διακριτική μεταχείριση και εις αυτών που δεν έχουν χρήματα. Για να υπάρχει καλή νομική λοιπόν ε, αρρωγή πρέπει να διακριθούμε το δικαίωμα αυτό με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το δικαίωμα της νομικής αρρωγής. Είναι μια πολύ σωστή αρχή και σχετική αρχή, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην έχει αρνητικές συνέπειες. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετική νομική βάση, διαφορετικά δικονομικά δικαιώματα. Και εάν προσπαθούμε να εισαγάγουμε κάτι ενιαίο, τότε υπάρχουν, να μην ξεχνάμε, χώρες ε, οι οποίες έχουν μια πολύ καλή νομική βάση και δεν πρέπει να επιδεινώσουμε την κατάσταση προσπαθώντας να εισαγάγουμε κάτι ευρωπαϊκό, κάτι ενιαίο. Και φυσικά έχω αντίληψη αυτού του κινδύνου και γνωρίζω πως ε, έχουν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με το κόστος και ξέρω πως αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως δεν το αρνούμε αυτό. Υπάρχουν ορισμένε ε, χώρε, όπω το Βέλγιο, για παράδειγμα, που αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε και προσπαθούν φυσικά να ε, κάνουν εξοικονόμηση πόρων Γι' αυτό και γίνονται περικοπές. Όμως εδώ πρόκειται για τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων και το θέμα δεν πρέπει να είναι το κόστος, αλλά πρέπει να είναι η δικαιοσύνη. Χρειάζεται διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβαση σε έναν καλό δικηγόρο και εδώ χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Στην οδηγία ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί πότε θα ε, γίνεται η χρήση της νομικής αρρωγής στην αρχή ή αργότερα. Επίσης, δεν έχω καταλάβει ποια είναι η αρμόδια αρχή, η αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της νομικής αρρωγής. Είναι κάποια εθνική υπηρεσία ή η υπηρεσία της ε, χώρας στην οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος. Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν έχουν διευκρινιστεί. Θεωρώ επίση ότι πρέπει να μιλήσουμε για το κόστος, για την ποιότητα της νομικής αρρωγής, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί, πρέπει να δοθούν εγγυήσεις για αυτή την ποιότητα. Πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε το κόστος. Στο Βέλγιο ασκούμενους στέλνουν να υπερασπιστούν αυτούς τους ανθρώπους δωρεάν. Όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και αυτή δεν είναι καλή αρχή. Υπάρχει στις κάτω χώρες επίσης ένα δικηγορικό γραφείο το οποίο ε, δίνει αποκλειστικά και μόνο δωρεάν ε, νομικές συμβουλές και νομική αρρωγή και χρηματοδοτείται από το κράτος. Ούτε αυτό όμως είναι και απόλυτα υγιές, διότι η νομική αρρωγή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή ισορροπία και μια καλή σχέση ανάμεσα στις, ε, στα δικηγορικά γραφεία και σε αυτή τη δωρεάν νομική αρρωγή. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια καλή ισορροπία, όχι μόνο το κράτος, όχι μόνο ασκούμενοι δικηγόροι, Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να διευκρινιστούν, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ψηλά ο πύχης της ποιότητας για τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Thank Σας ευχαριστώ. Τα μέλη της Επιτροπής νομίζω δεν θέλουν πια το λόγο. Ας ε, δώσω την ευκαιρία στην, ε, στους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου να τοποθετηθούν. Γιωχάννα Έγκστρομ από πλευράς Επιτροπής. Ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε το σχέδιο του εισηγητή, το διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε, είναι εξαιρετική η δουλειά που έκανε. Εμείς παρουσιάσαμε δύο εργαλεία για την νομική αρρωγή, μια οδηγία και μια σύσταση όπως ακούσαμε στην οδηγία εστιάσαμε στα επίγοντα ζητήματα και στη σύσταση ασχολούμασταν με τις υπόλοιπες χρήσεις. Αυτό έγινε για λόγους αναλογικότητας και επικουρικότητας. Όπως είπαμε, όλα τα ζητήματα έχουν τη σημασία τους. Θέλαμε όμως να αρχίσουμε να νομοθετούμε για τα σημεία που θεωρούμε εμείς ως πιο ενδιαφέροντα. Ε, παροχή νομικής αρρωγής ε, για τα πλέον ευάλωτα άτομα, δηλαδή αυτά που κρατούνται. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ενός δικηγόρου. Επίσης, ε, επεκτάθηκε η υπηρεσία σε όλους τους κατηγορουμένους και σε όλους τους υπόπτους στη δική σας πρόταση. Ας το συζητήσουμε. Όμως αυτοί που κρατούνται είναι σε πιο επισφαλή θέση, σε πιο ευάλωτη θέση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι αν διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή δεν θα υπονομευθεί το δικαίωμα αυτού του ανθρώπου να έχουν πρόσβαση στην νομική αρρωγή. Επίση, προτείνατε κριτήρια επιλεξιμότητα. Καλωσορίζουμε αυτό το βήμα και την πρότασή σας και είμαστε ανοιχτοί για να το συζητήσουμε. Μπορείτε να βρείτε κάτι αντίστοιχο στη σύστασή μας και θεωρούμε ότι είναι προσθέμενη αξία το να έχουμε μια σύγκληση και ισότιμους όρους μέσα από αυτήν την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, η ποιότητα της υπηρεσίας άλλο ένα ζήτημα που ευχαρίστως να συζητήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να το πραγματευτούμε στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία. βλέπουμε, στην επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και από κοινού νομίζω ελπίζουμε θα μπορέσουμε με αναλογικότητα να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για παροχή νομικής ε, αρρωγής στους κατηγορουμένους και στους υπόπτους στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών. Κύριος θα ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκα Ντεματές από πλευράς του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εκ μέρους του Συμβουλίου να ευχαριστήσω ειλικρινώς την εισηγήτρια για αυτήν την πρώτη εκδοχή εγγράφου που σκοπό έχει να μας δώσει τη θέση του Κοινοβουλίου για αυτήν την τόσο σημαντική ειδικία επί της οποίας μου επιτρέπω να το σημειώσω το Συμβούλιο και η Ιταλική Προεδρία έχουν καταβάλει σημαντικές διαπραγματευτικές προσπάθειες επειδή είναι και ένα από τα εργαλεία που προκύπτουν την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο του 2013 και για την προστασία των ε, ανηλίκων και τα δικαιώματά τους, αλλά και το τεκμήριο της αθωότητας. Θα αρχίσουμε να διπλωματευόμαστε για αυτά όταν το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο. Όπως υπόθηκε, ε, την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου συζήτησε το θέμα αυτό ξανά και ξανά. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και μια σειρά από τις αρχές ε, που αναφέρονται στην οδηγία ήδη έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κατών μελών. Βεβαίως η συμφωνία δεν ήταν ακόμα συνολική, διότι υπάρχουν κάποιες θέσεις που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Έγινε κάποια αναφορά στο τερισμένη πτυχές της οδηγίας, πώς προς το σκοπό όλοι συμμεριζόμαστε, σημειώνει ότι σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγο πολύ υπάρχει το σύστημα της νομικής αρρωγής του Legal Aid. Οπότε είναι απαραίτητο οι κανόνες της οδηγίας αυτής να μπορούν να συμπληρώσουν όπως πρέπει τα συστήματα που ήδη υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια ανάγκη ισορροπίας την οποία πρέπει να σεβαστούμε και το θέμα δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά μέσα, αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρονται. Από την άποψη αυτή, το Συμβούλιο σημειώνει με ενδιαφέρον τις διάφορε ιδέε τη έκθεση. Θα τι αξιολογήσει και θα φροντίσουμε να έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο για να περάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από την πλευρά λοιπόν του Συμβουλίου δεν μπορώ παρά συμπαραταχθώ με όσα είπε η κυρία Ζίπελ. Ε, εργαστήκαμε σε μια πρόταση της Κομισιόν που από την αρχή είχε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, πολύ αυστηρό. Και ίσως Δεν ήταν ε, και ακριβώς ε, η σύσταση που είχε δώσει το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 για ένα συνολικό σύστημα Legal Aid. Η πρόταση που έχουμε στα χέρια μας και την οποία επεξεργάζεται το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τις ιδέες του Κοινοβουλίου. Απλώς να σημειώσω ότι οι ιδέες αυτές επειδή θα πρέπει να φτάσει σε ψηλότερο επίπεδο η οδηγία αυτή από όσο είχε αρχικά στοχεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σημειώσω ότι η πρόταση αυτή έχει διαφορετικό λόγο ύπαρξη, με πολύ πιο περιορισμένη μελέτη αντικτύπου σε σχέση με τι προτάσει που εδώ γίνονται από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Ε, σημειώνει το γεγονό ότι για την πρόταση αυτή τα εθνικά κοινοβούλια έχουν εκφράσει την άποψή του ω προ την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Να συμφωνήσω με το αίτημα που ακούστηκε στην αίθουσα αυτή, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πτυχέ αυτέ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όπω είπα όμω, Αναμένουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο θα φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ωστόσο πιο σύντομα ε, να φτάσουμε σε μια δυνατή λύση. Thank you very much. Um, Ευχαριστούμε πολύ και τώρα να δώσω το λόγο πάλι στην... στον εισηγητή για να ε, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους και τους εισηγητές που πήραν το λόγο. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνονται αρκετά διαλλακτικοί και ανοιχτοί στην προσέγγιση τους. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Κοινοβούλιο με τους χιώδεις εισηγητές, θα μπορέσουμε να έχουμε, μια, ε, θα, να έχουμε αρμονικές διπλωματεύσεις και με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Να αντιδράσω στις παρεμβάσεις που άκουσα να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Σαρχεντίνη για την κατάσταση στην Ολλανδία. Βλέπουμε από τη μια ε, το κόστος των δικών να φτάνει στα ύψη και από την άλλη να υπάρχει όλο και λιγότερη νομική αρρωγή. Υπάρχει εδώ ε, μια αντίφαση σε κοινωνικό επίπεδο. Ε, δηλαδή, εάν υπάρχει, αν κανείς είναι πλούσιος, μπορεί να πληρώσει και ένα καλό συνήγορο, οπότε ενδεχομένως να μειώσει και την ποινή του. Και αν κάποιος δεν έχει λεφτά, θα έχει αυστηρότερη ποινή γιατί δεν είχε καλή υπεράσπιση. Ε, πρέπει να φροντίσουμε η πρόσβαση στο δικαίωμα αυτό να είναι εγγυημένη για όλους. Είμαι ιδιαίτερα ανοιχτό για να συζητήσουμε και το θέμα των ανηλίκων. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δύσκολο. Θα ήθελα να προβλέψουμε αυτομάτως το ακέραιο δικαίωμα και των παιδιών ε, σε πρόσβαση στην νομική ρογή. Όμως στην οδηγία για τα δικαιώματα των ανηλίκων νομίζω ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Εμείς θα πρέπει να επιδιώξουμε να διοργανώσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών νομοθετημάτων και είμαι σε και έχω την ε, απόλυτη διάθεση να το κάνω. Το ΕΛΚ μιλά για την αναλογικότητα και καταλαβαίνω ότι ε, σε τι αναφέρονται. Όμως η πρόσβαση στο δικαίωμα της υπεράσπισης δεν μπορεί να μετράται με όρους αναλογικότητας. Ε, δεν ανέφερα αριθμητικά στοιχεία, ούτε για να φτάσουμε σε μειωματική και πλήρη εναρμόνιση της νομικής αρρωγής. Αυτό που θα ήθελα είναι να υπάρχει μια ε, εξελαχίστων τουλάχιστον βάση για να ε, είναι εγγυημένο το δικαίωμα και ως προς την διαδικασία νομίζω μπορούμε να συναντηθούμε με το Σκιώδης για να ετοιμάσουμε τις τροπολογίες, εάν χρειαστούν διευκρίνηση από πλευράς μου ευχαρίστως. Απλώς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι τροπολογίες αυτές υποβληθούν. Μπορούμε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση όπου όλοι να αισθάνονται ότι καλύπτονται σε αυτή την Επιτροπή. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση για να έχουμε και αποτελεσματικές διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να φτάσουμε σε μια κοινή θέση με τους σκιώδες εισηγητές δυνατόν και ελπίζω να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Εμείς σας ευχαριστούμε. Για την κατάθεση τροπολογιών έχουμε ορίσει τη 13η Ιανουαρίου στις 12 ως προθεσμία. Για το επόμενο σημείο, ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Αλφάνο, ε, αρμόδιο για τι εσωτερικέ υποθέσει και τον κύριο Ορλάντο για τη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, διότι ακόμη δεν έχουν έρθει. Στις παραδέκα ε, θα συνεχίσουμε. Μπορείτε να πιείτε ένα καφέ ή ό,τι θέλετε να κάνετε. Να 50.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

Uh, Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Εάν θέλετε να καθίσετε Remaining members to... και να ζητήσω από τους συναδέλφους που έμειναν στην αίθουσα να παρακολουθήσουν. We have Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ορλάντο, Υπουργό Δικαιοσύνης, και εάν όλα πάνε καλά αργότερα και με τον κύριο Αλφάνο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και θα συζητήσουμε για τα συμπεράσματα για την έκβαση της Ιταλικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών. Να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Ανδρέα Ορλάντο, Ιταλό Υπουργό Δικαιοσύνη, που θα μας παρουσιάσει τις δραστηριότητε της Ιταλική Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Ο κύριος Αλφάνο που θα έρθει αργότερα αν όλα πάνε καλά. Πρόσφατα πήρε μέρος στην ε, υπουργική συνάντηση Υπουργών Εσωτερικών στο Παρίσι G6. Θα μας μιλήσει λοιπόν για τις εσωτερικές υποθέσεις και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να μας απαντήσει όλες σε ερωτήσεις που ενδεχομένω θα έχουμε αργότερα, εφόσον έρθει, ως προς την προκτική διοργάνωση της συζήτησης. Επειδή έχουμε εδώ μόνο τον κύριο Ορλάντο, θα ξεκινήσουμε μαζί του και μετά οι συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο. Κύριε Ορλάντο, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Άλμπρεχτ, ευχαριστώ μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που με προσκαλέσατε και για να σας αναφέρουμε το έργο μας κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης φτάνει στο τέλος της. Οπότε ήθελα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα που είχαμε στο τελευταίο εξάμεινο στον τομέα αρμοδιοτήτων μου. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ικανοποίηση ότι καταφέραμε να τηρήσουμε τι υποσχέσει μα, ακόμη και ενώπιον αυτή τη επιτροπή, κατά τη διάρκεια τη αρχική ακρόαση που είχαμε τον περασμένο Ιούλιο. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου σε όλους τους τομείς δράσης μας. Από την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα του δικαιώματος προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων μέχρι την ε, αστική και ποινική συνεργασία αλλά και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, την εκπαίδευση δικαστικών, βασικό στοιχείο της ε, οικοδόμησης αμοιβές εμπιστοσύνης για τις διάφορες νομοθεσίες και τους λειτουργούς του δικαστικού συστήματο. Τώρα θα ήθελα να παρουσιάσω ανακεφαλαιωτικά τα βασικά συμπεράσματα, της, τα βασικά αποτελέσματα τη Ιταλική προεδρία στον τομέα αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή σα και μετά να εμβαθύνουμε αν θέλετε βάσει των ερωτήσεών σα. Ο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων ε, έτυχε έντονη διαπραγματευτική δραστηριότητα το τελευταίο εξάμεινο, παρόλο που υπήρχαν πολλά νομικά εμπόδια και θέματα αρχή λόγου χάρη θέματα που είχαν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την επικουρικότητα. Από το Συμβούλιο πετύχαμε να έχουμε την τελική έγκριση και επίλυση ενός προβλήματος που είχε προκύψει στην αρχή των διαπραγματεύσεων για τη συμπερίληψη των ε, δεδομένων στον δημόσιο τομέα και στο πεδίο ισχύω του ε, κανονισμού. Μετά το άτυπο συμβούλιο του Μιλάνου μπορέσαμε να πετύχουμε, να συμπεριλάβουμε στον κανονισμό κανόνες που δίνουν στα κράτη-μέλη ε, επαρκέ περιθώριο ευελιξίας για την ε, μεταχείριση και την επεξεργασία δεδομένων στον δημόσιο τομέα βάσει των ειδικών απαιτήσεων που υπήρχαν σε αυτό τομέα. Αυτές οι, ε, αυτοί οι κανόνες δεν αλλάζουν την ουσία του κανονισμού που διαφυλάχθηκε. Όμως ε, η μεγαλύτερη ευελιξία για να προστατευτούν οι εθνικοί ε, ειδικοί νόμοι σε αυτόν τον τομέα έχει προβλεφθεί. Και υπάρχει και ένα επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που είναι συμβατό με το επίπεδο προστασίας όπως το προβλέπει ο κανονισμός. Επιπλέον, καταφέραμε να έχουμε μια προκαταρκτική συμφωνία στο Συμβούλιο για τους κανόνες τέταρτου κεφαλαίου του κανονισμού. Το κεφάλαιο που αφορά τις υποχρεώσεις των υπευθύνων και των φορέων που ε, επεξεργάζονται τα δεδομένα. Το κεφάλαιο αυτό είναι καθοριστική σημασίας για τους οικονομικούς φορείς που στη δράση τους ε, μπορεί να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Ορίζονται πρότυπα που θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στη δραστηριότητα επεξεργασία δεδομένων και έτσι θα προσφέρει ισορροπία στο υψηλό επίπεδο προστασία των δεδομένων και τον περιορισμό του διοικητικού άχθους για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες ώστε να υπάρχουν οι σωστέ συμπεριφορέ, χωρί όμω ασφικτικά να πιεστεί η πρωτοβουλία των ιδιωτών. Πιστεύουμε ότι καταφέραμε να έχουμε εδώ μια ικανοποιητική συμβαστική λύση. Τέλο, στο Συμβούλιο Τζάι τη 4η Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί στήριξαν το γενικό αρχιτεκτόνημα μια πρόταση ε, για να επιληθεί το θέμα που και αυτό έχει συζητηθεί από πολύ καιρό, για την ενιαία θηρίδα για τις επιχειρήσεις, το λεγόμενο one-stop shop, πρόταση της Προεδρίας και αυτή, η οποία σκοπό έχει να διατηρήσει το στόχο απλούστευσης και συνέπειας στην εφαρμογή του κανονισμού, όπως προκύπτουν από την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ταυτόχρονα προβλέπεται ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία για του πολίτε βάσει του κριτηρίου εγκύτητα και τη πρόσβαση σε ένδικα ε, και ένδικα διοικητικά ε, μέσα. Εφόσον υπάρξουν παραβιάσει των δικαιωμάτων που έχουν σχέση με τον ιδιωτικό βίο. Οι υπουργοί συμφώνησαν, οπότε θα υπάρξει και περαιτέρω τεχνική επεξεργασία του θέματος για να μεταφραστεί και σε λεπτομερέστερους κανόνες. Η Προεδρία δεν παραμέλησε επίσης την οδηγία για τις ποινικέ διοικητικές διαδικασίες και τις αστυνομικές δραστηριότητες, θεωρώντας ότι χρειάζεται μια συνεπής και συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των δύο νομοθετημάτων και για να έχουμε το μέγιστο επίπεδο ε, προστασίας μαζί με την ε, αποτελεσματική ε, δικονομική εξέταση του θέματος. Στο πεδίο της οδηγίας η διεθνής ε, ανταλλαγή δεδομένων ε, ήταν κάτι που συζητήθηκε, όμως δεν ήταν ακόμη όριμη η συζήτηση για να καταλήξουμε σε συμφωνία και επειδή υπάρχουν πολλά σημεία επαφής με τον γενικότερο κανονισμό που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το συγκεκριμένο ντοστιά. Από τη δική μα την πλευρά μπορούμε απλώς να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι από τον Ιούνιο εφέτος, κάθε φορά που συνήλθε το Συμβούλιο Τζάι, προέκυψε τουλάχιστον μια συμφωνία για ένα θεμελιώδης τμήμα του νομοθετήματο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο με ταχύ ρυθμούς προχωρά προς την έγκριση μια συνολική συμφωνία για το κείμενο, ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει τη συναπόφαση. Στον ποινικό τομέα έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία και για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και στην Αθήνα ε, υποσχεθήκαμε μία λύση ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους Ευρωπαίους πολίτες στα ίδια ένδικα μέσα με τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ίσως ε, να χρειαστεί αλλαγή στο εσωτερικό νομικό μας πλαίσιο, διότι οι εθνικές νομοθεσίες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την αλλαγή για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στην ε, στους κανόνες που προέκυψαν. Τώρα στον ποινικό τομέα δώσαμε μεγάλη ε, έμφαση στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και την θέση του, ε, ένα σημαντικό στοιχείο του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης. Σε σχέση με τις ανακριτικές ε, δυνατότητες του της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και την κατανομή αρμοδιοτήτων με τα κρατικά υπουργεία, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων των ε, υπόπτων και των προσαχθέντων, μπορέσαμε να δώσουμε ένα γενικό προσανατολισμό. Ένα γενικό προσανατολισμό ώστε να υπάρχει και ένας βαθμός ανεξαρτησίας στα μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δικαιώματα διερεύνησης και ανάκρισης ιδιαίτερα προηγμένα. Η τεχνική πτυχή του θέματος αυτού θα οδηγήσει στους λεπτομερείς κανόνες στον όλο τομέα και ελπίζουμε να υπάρξουν αποφασιστικά βήματα πρόοδου με την επόμενη Προεδρία προκειμένου να υπάρξει και συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών πρωτοβουλειών στον ποινικό τομέα, η Προεδρία ξεκίνησε τι διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο ω προ την οδηγία για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων τη Ένωση. Σε πολύ σύντομο χρόνο είχαμε εξωσημείωτη πρόοδο προς ένα ε, συμπεφωνημένο κείμενο. Λίγα είναι τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει αίσια έκβαση σύντομα με την επόμενη Προεδρία. Θέλουμε να τονίσουμε και τη σημαντική πρόοδο στην διαδικασία μεταρρύθμισης της Eurojust. Η Προεδρία υπέβαλε στους υπουργούς μια μερική γενική προσέγγιση για το κείμενο που αφορά τις εξαιρέσεις για την προστασία των δεδομένων και θα χρειαστεί βεβαίως και περαιτέρω τεχνική επεξεργασία αλλά και για τις προδιαγραφές της μελλοντικής ευρωπαϊκής εισαγγελίας καθώς το επίπεδο πρόοδου των δύο ντοσχέ είναι διαφορετικό αλλά μπορούμε από κοινού να φτάσουμε σε κοινό πλαίσιο και για την πρόταση αυτή. Το Συμβούλιο σύντομα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο αναζητώντας μια κοινή ε, θέση και να προκειμένου να υπάρξει ταχεία έγκριση του κανονισμού ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων ή των κατηγορουμένων στις ποινικέ διαδικασίες έχει ξεκινήσει εξετός του θέματος στο Συμβούλιο βάσει των όσων προβλέπονται για το τεκμήριο αθότητας και προκειμένου να υπάρξει μια γενική τοποθέτηση στο Συμβούλιο Τζάι του Δεκεμβρίου. Με μεγάλη χαρά ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσει στη διαδικασία της συναπόφασης με τα μέλη της Επιτροπής σας και ε, πολύ σύντομα θα γίνει κάτι τέτοιο με ιδιαίτερες με ιδιαίτερη πρόοδο σε όσα έχουν να κάνουν και με την νομική αρρωγή, legal aid. Αν και υπάρχουν ακόμη ζητήματα σε εκκρεμότητα που θα πρέπει να ετοιμαστούν από τις ανάλογες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου ως προς την αντιμετώπιση των σοβαρών μορφών εγκλήματος όπως οι, οι διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις ή εμπορία ανθρώπων θα υπάρξει διαρκή συνεργασία μεταξύ Προεδρίας και κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και της ε, κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η πολιτική πρό, πρόκληση. Διότι οι εγκληματίε και οι εγκληματικέ οργανώσει δεν θα πρέπει να έχουν έσοδα κανενό είδου και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν από τι παράνομε δραστηριότητέ του και με οποιαδήποτε τρόπο και αν τα έχουν αποκτήσει. Σε αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και έτσι η Προεδρία ε, έδωσε ε, συνέχεια στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, καθώς και οργάνωσε μια εντελεχή συζήτηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι μορφές δίμευσης ή κατάσχεση βάσει δικαστικών αποφάσεων εντός και εκτός των ποινικών διαδικασιών με, ένα υψηλό, ε, επίπεδο, με μια υψηλού επίπεδο εκδήλωση που οργανώθηκε στη Σιρακούσα 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Ε, τα θέματα αυτά τα εξέτασαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνη στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου και ελπίζουμε ότι θα οδηγήσουν στι επόμενε νομοθετικέ πρωτοβουλίε για το όλο θέμα. Όπω ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, η Ιταλική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα τη εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών στα κρατικά υπουργεία. Γι' αυτό προτείναμε στους Υπουργούς ένα κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που καθορίζει τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες σε αυτό το χώρο, καλώντας όλους τους ε, ε, συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τις σχολές και τους οργανισμούς εκπαίδευσης, τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσφέρουν ε, δυνατότητες εκπαίδευσης και ανταλλαγής εκπαιδευτικών συστημάτων μεταξύ των δικαστικών αρχών. Τέτοια, αυτά τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο Τζάι του Δεκεμβρίου. Ε, μια επίση πλούσια συζήτηση είχαμε με τα κάτι μελη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα θέματα αρμοδιότητα στην ποινική δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, αλλοδαπών μαχητών. Προωθήσαμε για αυτό το σκοπό ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών ε, Δικαιοσύνη, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Eurojust και του συντονιστή για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία ώστε να ορίσουμε σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό τις ανάλογες αποκρίσεις στις εκκλήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να υπάρξει ένα ισχυρό πλαίσιο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προφανώς την όλη αυτή συζήτηση εντάσσεται και το θέμα που εξέτασαν οι συνάδελφοι των εσωτερικών ε, υποθέσεων για να δούμε πώς η αποτροπή μπορεί να λειτουργήσει ως έννοια παράλληλα με τη δική μας ε, δράση. Τα Υπουργεία Εσωτερικών ασχολούνται λοιπόν με το πώς μπορεί να παρέμβει κανείς στο όλο φαινόμενο κατά τη διάρκεια ενώ εμείς στο Υπουργείο Δικαιοσύνη ασχολούμαστε με την πρόληψη και την ε, επιβολή ποινών στο φαινόμενο αυτό, ακόμη και με μορφές εκτέλεσης της ποινή που λαμβάνουν υπόψη της ιδιαιτερότητας του φαινομένου των αλλοδαπών μαθητών. Ε, εν είδη συμπεράσματος, να πω στα μέλη της Επιτροπής σας ότι η Ιταλική Προεδρία απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Τζάι του Δεκεμβρίου για να καλέσει τα κατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν συνέχεια στην απόφαση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κρίμ στην προηγούμενη θητεία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η διαφθορά και, τη διαφθορά και την ε, ανακύκλωση παράνομων προσόδων. Ε, υπήρξαν ενδιαφέρουσε ιδέες εδώ και στο τεχνικό και στο διαδικαστικό επίπεδο. Στον πρόεδρο της Επιτροπής θέλω να πω ότι η Προεδρία μας υπέβαλε στο Συμβούλιο ε, των ε, Υπουργών νέα στοιχεία για το θέμα αυτό. Επίσης, έναν υπενιγμό να κάνω για τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που είχε η Ιταλική Προεδρία στο χώρο του αστικού δικαίου. Θα ενημερώσουμε αναλόγω τον ε, πρόεδρο Βόμποντα, αλλά θέλω να ενημερώσω και την Επιτροπή σα ότι η συμφωνία που πετυχώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τι διαδικασίε ε, αφαιρετικότητα ή πτώχευση είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, ιδίω αυτού του καιρού οικονομική κρίση. Είναι σημαντικό για την επιβίωση των επιχειρήσεων, στι οποίε θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία εφόσον εγκριθεί αυτή η διαδικασία. Εδώ εμπλέκονται και προφανές, προφανείς νομικής νομικές επιπτώσεις γιατί η κρίση όπως ξέρουμε έδωσε πολλά ενάυσματα στο οργανωμένο έγκλημα και στα παράνομα έσοδα των εγκληματιών έδωσε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και η έλλειψη μιας διαφανούς διαδικασίας πτώχευσης δημιούργησε πολύ επικίνδυνε συνθήκε για τι επιχειρήσει που είχαν πληγεί από την ε, κρίση. Επίση, μια γενική προσέγγιση για κάποια αμφιλεγόμενα θέματα ήδη ε, έχει προβλεφθεί, αλλά τη συνέχεια θα δώσει η Λετωνική Προεδρία στι διαπραγματεύσει με το Ευρωκοινοβούλιο. Επίση, πρόοδο επιτεύχθηκε στο θέμα για την απλούστευση και την αποδοχή κάποιων δημόσιων εγγράφων. Υπήρξε συνένεση στο Συμβούλιο για κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ που έχουν να κάνουν με τα βασικά σημεία τη πρόταση κανονισμού. Εν τέλει, δώσαμε νέα αίθουσα στην πρόταση κανονισμού για το καθεστώς το κληρονομικό σε περίπτωση γάμων και και συμφώνων συμβίωση. Υπήρξαν δυσκολίε στο Συμβούλιο, εσωτερικέ δυσκολίε, για να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση, αλλά προχωρήσαμε. Τέλος, να επισημάνω στην Επιτροπή σας ότι η Ιταλική Προεδρία Εν είδη συμπεράσματος, η Ιταλική Προεδρία ε, λειτουργήσε σε ένα θεσμικό πλαίσιο σε κατάσταση μεταβολής και είδε και κατάφερε να οριστούν νέοι στρατηγικοί προσανατολισμοί παρόλα αυτά στον τομέα ασφάλειας και δικαιοσύνης. Υπ' αυτές τις συνθήκες ελπίζουμε ότι ε, υπηρετήσαμε σωστά το σκοπό της ενίσχυσης του, του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών με αυτές τις ε, σημειώσεις και παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστούμε. Ήσασταν ε, πληρέστατος. Ο κύριος Αλφάνο δεν έχει καταφτάσει, είναι καθοδόν. Θα αρχίσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων ε, για τον κύριο Ορλάντο. Ο κύριος Μπούνι θα αρχίσει και ακολουθούν άλλοι τρεις. Μποντ, ο κύριος Μποντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Ήταν ξεκάθαρη παρουσίασή σας. Ευχαριστώ τον, την Ιταλική Προεδρία για τη συμβολή της. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμήσει κανείς την ουσιαστική εισφορά της ε, Ιταλικής Προεδρίας. Για τον κανονισμό, τώρα για την προστασία ατομικών δεδομένων, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Έχω την εντύπωση πως είστε υπερβολικά αισιόδοξο. Και βλέπετε υπερβολικά θετικά τα επιτεύγματα. που σημειώθηκαν μέχρι σήμερα και ως προς τις προβλέψεις σας για την ε, τελική έγκριση μετά την ε, και τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Μιλήσατε για την ενιαία θηρίδα, One Stop Shop. Η λύση που εξετάζεται απέχει πόρο από την αρχή, δηλαδή ένα ενιαίο σημείο επαφής Δεν νομίζω ότι γίνεται σεβαστή αυτή η αρχή στον κανονισμό. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει συμφωνία των κρατών μελών για την ενιαία θηρίδα. Πώς βλέπετε αυτό το θέμα. Επίσης, οι λύσεις στις οποίες θα καταλήξουμε θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες. Οι εξαιρετικά περίπλοκες λύσεις που προτάθηκαν για την ενία θηρίδα νομίζω θα δημιουργήσουν μεγάλες δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους. Κλείνοντας να σε ευχαριστήσω και πάλι για την... θα ε, σας καταφέρατε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Αν θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την ενία θηρίδα θα το εκτιμούσαμε, διότι έτσι θα μας διαφωτίσετε για τη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπον. Τσινίτσι, τώρα παρακαλώ να περιοριστείτε ε, στα δύο λεπτά στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για την ε, πληρέστατη παρουσίαση των θεμάτων που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Πρόκειται για μια δουλειά ε, ιδιαίτερα σημαντική για θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Θέματα που ε, απασχολούν καθημερινά την Επιτροπή μας. Ο Υπουργός ανέφερε τα βασικά νομοθετήματα όπου έγιναν κάποια σημαντικά βήματα πρόοδου. Όλος ιδιαίτερος Πρέπει να πω ότι παρακολούθησα τον κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Υπουργό είπε ότι εδώ πρέπει να και ξεκίνησε να γίνεται προσπάθεια για τον ρυθμό των αρμοδιοτήτων. Εδώ όμως πρέπει να φροντίσουμε να διαχωρίσουμε σωστά το τι κάνουν άλλοι υπάρχοντες οργανισμοί όπως η Eurojust, η Europol και, και η Όλαφ σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε και να φροντίσουμε να υπάρξει ένα ε, σωστό ε, ορισμό των μεν και των δε. Επίση, αρκετή δουλειά έγινε για να προχωρήσουν οι δύο προτάσει οδηγία για το τεκμήριο οθετία ε, αθότητα και την νομική αρρωγή. Εδώ, Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα για το τι διαχωρισμό αρμοδιοτήτων θα υπάρξει μεταξύ των οργανισμών που ανέφερα και τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είμαι πεπισμένη ότι οι δικονομικέ εγγύησει τι οποίε προβλέπετε με τι δύο προτάσει οδηγίε που ανέφερα, αυτέ οι δικονομικέ εγγύησει είναι πολύ σημαντικέ για την όλη πρόταση, την πρόταση και για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάκρισης και την ε, εκδίκαση των υποθέσεων όπως θα προκύπτουν εξαιτία της δράσης αυτής της υπηρεσίας. Ε, να σας ευχαριστήσω και όλας Υπουργέ γιατί μιλήσατε και για την δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της εργασίας της Υποεπιτροπής ΚΡΙΜ και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες τις ε, μορφές. Ξέρουμε ότι με τη δράση της το οργανωμένο έγκλημα τελικά επιβαρύνει σημαντικά την πραγματική οικονομία όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Ευχαριστούμε λοιπόν Υπουργέ και θα θέλαμε λίγο να εμβαθύνετε στα θέματα για τα οποία σας έθεσα ερωτήσεις. Thank you, Ευχαριστούμε κυρία Τσινίτση. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Ευχαριστούμε κύριο Λάντο. Ε, εξεργαστήκατε την οδηγία για την εφαρμογή της αρχής μεταχείρισης για όλους ε, ανεξαρτήτως ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκεύματος, εθνοτικής προέλευσης, ε, της ε, για την ισότιμη μεταχείριση. Και μιλήσατε για τα, την ελευθερία σύναψης ε, συμβάσεων ε, ως προς το αστικό δίκαιο. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό θα απλήξει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, ε, άλλοι παραπονιούνται ότι είναι ασαφέστατη η διατύπωση και αν εγκριθεί το νομοθέτημα θα οδηγήσει σε απεκτές ερμηνείες των διατάξεων. Μη κυβερνητικέ οργανώσει από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο Γιούγκερ ζητώντας αναδιατύπωση για να μην δημιουργηθεί η πολιτική ανακολουθία λόγω της εφαρμογής ε, του νομοθετήματος. Εσείς τι προτείνετε ε, στη Λετωνική Προεδρία για αυτήν την οδηγία. Άλπρες. Ε, ευχαριστώ. Έχουμε και άλλους άλλα μέλη που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Παρακαλώ να είστε σύντομοι για να ακούσουμε τις απαντήσεις και να περάσουμε και στον κύριο Αλφάνα. Αλφάνο που μόλις ήρθε. Ε, η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας Υπουργέ Ορλάντο. Καλημέρα σας Υπουργέ Αλφάνο. Χθε γιορτάσαμε την Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ξέρουμε πως αυτό απασχολεί όλη την Ευρώπη πολύ σοβαρά ήδη το 2013 και μετά το 2014 με ιδιαίτερη ένταση ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμένου το Συμβούλιο ζήτησε από την Ιταλία να ενισχύσει τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς. Ιδίω για την αναθεώρηση των όρων παραγραφής που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ε, ελαφρύ, ελαφρύς. Σας ζητώ λοιπόν να μου πείτε αν στην Ιταλία έγινε προσπάθεια να ακολουθήσουμε τις ευρωπαϊκές επιταγές και στην Ευρώπη ποια ήταν τα συγκεκριμένα μέτρα που προωθήθηκαν για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδηγία για την ε, διακριτική μεταχείριση equal treatment και αυτά που είπε προηγουμένως και ο συνάδελφο, Σας ζητώ να μου πείτε τι ε, εξελίξει υπήρξαν στο Συμβούλιο. Είχαμε επιμείνει στην ενισχυμένη συνεργασία για να ξεπεράσουμε το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η οδηγία αυτή. Ήταν απογοητευτικό το αποτέλεσμα όμως, δεδομένου του τόσο ευαίσθητου ζητήματος που καλύπτει η οδηγία αυτή. Καλό θα ήταν να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο, αλλά κυρίω το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα των κρατουμένων. Στην παρουσίαση του προγράμματο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είχε γίνει λόγο για την ανταλλαγή των πρακτικών και την αμοιβή αναγνώριση των ποινών ή την ε, προσωρινή αναστολή. Ω προ αυτά, τι έγιναν, τι έγινε για τα δικαιώματα των κρατουμένων στα πλαίσια τη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ε, διαχείριση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, αλλά και για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένα ενίο νομικό πλαίσιο για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλα τα κράτη-μέλη μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδηγία την οδηγία για την καταπολέμηση του δημοσιονομικού εγκλήματος Η οδηγία αυτή ξέρουμε ότι θα αποτελέσει τη βάση για την ίδρυση του, ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι πρόοδος επιτεύθηκε σχετικά και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της δράσης της Επιτροπής Κρίμα από την προηγούμενη θητεία. Είναι σημαντικό η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα να καταπολεμηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζουμε ότι η σχετική δράση θα προχωρήσει. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. ξεχνάτε και τους διερμηνείς, λέει γενικά ο Πρόεδρος. Μιλάτε υπερβολικά γρήγορα. Κύριε Βάνου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Υπουργό Ορλάντο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που έκανε. Μίλησε για του ξένου μαχητέ και μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την ειρήνη στον κόσμο. Κυρίως στη χώρα μου βλέπουμε σαφέστερε εκδηλώσει αυτού του φαινομένου χρειάζονται αποτρεπτικές ε, κυρώσεις ε, και θα ήθελα να ε, μας πείτε τι πιστεύετε σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 2028 για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Έχετε κάποια πρόταση σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Έχετε προθέσεις για την ανάληψη αποτρεπτικών κυρώσεων. Άμπρεχτ. Ευχαριστούμε. αυτέ είναι οι ερωτήσεις, το set ερωτήσεων προ τον κύριο Ορλάντο. Θα ήθελα να ακούσουμε κάποιες σύντομες απαντήσεις και μετά θα περάσουμε στον κύριο Αλφάν Παρακαλώ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις στο τμήμα που αφορούν την ε, Ιταλική Προεδρία και στο τι έγινε δηλαδή συγκεκριμένα στο Συμβούλιο και νομίζω ότι καλό θα ήταν να δοθούν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις στους βουλευτές για τα ε, θέματα που έθεσαν συνολικά, αλλά δεν είναι εδώ αυτή η κατάλληλη ευκαιρία, πιστεύω, για διεξοδικέ απαντήσεις. Για το One Stop Shop στην ενιαία φυρίδα οργανώσαμε μια συζήτηση προσανατολισμού το Δεκέμβριο. Η ομάδα εργασίας ελπίζουμε να βρει τεχνικές λύσεις για το θέμα αυτό, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Οι λύσει θα πρέπει να καλύπτουν από τη μια τη θέση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την άλλη της πλειοψηφίας των κρατών μελών Επ' αυτού Ο σκοπός είναι να υπάρχει πρόσβαση σε ένδικα μέσα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων ή μη σεβασμού της προστασίας των ε, δεδομένων στη χώρα προέλευσης, καταγωγής. Το θέμα για να βρεθεί μια λύση είναι ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συντονισμού. Εάν υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί λύση και μετά την άποψή μου, να πω πως πιστεύω ναι. Ε, μπορούμε να καλύψουμε αυτή την ε, ανησυχία που έχουν οι περισσότεροι, αλλά από γενική. Απόψη, κύριε Μποντ, μιλήσατε για μια υπέρμετρη αισιοδοξία. Όταν ξεκίνησε το εξάμεινο για το θέμα αυτό πρέπει να πω ότι ήμουν ιδιαίτερος απεσιόδοξος. Αν αυτή τη στιγμή ε, αν αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξο, είναι επειδή μερικά κομβικά σημεία κάπως επιλύθηκαν ε, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε και να αναφέρω ένα. Ξεκινήσαμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο με μεγάλη πόλωση μεταξύ των κρατών μελών, με δύο στρατόπεδα. Η ΜΕΝ στο νέο κανονισμό έβλεπαν τον κίνδυνο να Ε, καταστραφούν τα επιτεύγματα της εσωτερικής νομοθεσίας τους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι θα δημιουργηθεί υπερβολικό άχθος για τις επιχειρήσεις. ως προς τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονταν για να μεταφερθούν οι νέοι κανόνες. Νομίζω το κομβικό σημείο αυτό το επιλύσαμε με την ευελιξία που επέδειξαν όλοι, μπορέσαμε να ισορροπήσουμε τις διαφορετικές θέσεις. Και μπορούμε τώρα να ελπίζουμε σε σημαντικά βήματα πρόοδου. Αν δεν είχαμε επιλύσει αυτό το κομπικό σημείο, θα είχε μπλοκαριστεί η εξέλιξη του ντοσχέ. Γι' αυτό εξέφρασα την ικανοποίησή μου και δεν είναι καθόλου προπαγανδιστική η τοποθέτησή μου. Νομίζω ότι η επόμενη Προεδρία θα μπορέσει να ε, εργαστεί επειδή ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο και θα μπορέσει απρόσκοπτα να συνεχίσει τον ντοσχέ. Αυτό που είναι σημαντικό, το ανέφερα και στην παρουσίασή μου, είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, για ένα περίπλοκο πολιτικό πλαίσιο που θα, δεν θα μπορούσε να καλυφθεί σε ένα ολόκληρο εξάμεινο. Υπάρχουν εδώ πολιτικές ισορροπίες στις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή και άλλαξε και ο υπεύθυνο εξέταση του θέματος αυτού στην ε, κυβέρνηση Ομπάμα. Οπότε, αυτό ήταν και ένας αστάθμητος παράγοντας για την εξέλιξη του ΣΚΕ. Όμως, μπορούμε να πούμε ότι οι προποθέσει είναι ευνοϊκές για να προχωρήσουμε. Δεν ε, ξεκινήσαμε με τις ίδιες προϋποθέσεις πάντως στην αρχή του εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά το θέμα που έθεσε η κυρία Κινίτσι, νομίζω δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις. οι απαιτήσει επαγγελματισμού που προβλέπονται σήμερα θα γίνουν σεβαστέ. Θα ε, επεξεργαστούμε περαιτέρω τι σχέσει με, με του άλλου φορεί και του οργανισμού. Αλλά η ισορροπία στην οποία κατέληξαν τα κράτη-μέλη μεταφράζεται σε μια συμφωνία για την ε, ίδρυση τη Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις σχέσεις της με τις εθνικές. Εδώ τέθηκε και μια ερώτηση εύστοχη κατά την άποψή μου. Το βασικό πρόβλημα θα είναι το θέμα του ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων. Εδώ υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, πολύ μεγάλες. Προσπαθήσαμε να περάσει η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι αντιστάσεις πάρα πολλών κρατών μελών ήταν τεράστιες. Σε ό,τι λοιπόν αφορά το τι θα γίνει το ερχόμενο εξάμεινο, νομίζω ότι θα πρέπει έμφαση να δοθεί εκεί ακριβώς. Ως προς την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης για τα ερχόμενα χρόνια και το θέμα αυτό προβλέφθηκε ως θέμα προτεραιότητας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κράτησης, οργανώθηκαν συναντήσεις τεχνικού επίπεδου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και για το θέμα των σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Αλλά πιστεύω, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, ότι αυτό το ντοσχέ δεν ήταν το πιο ενδιαφέρον για τους άλλους, για τα κατημέλη στο εξάμεινο αυτό, γι' αυτό και δεν έτυχε της κατάλληλης προώθησης. Στο επόμενο εξάμεινο ελπίζουμε ότι θα το δουν με, περισσότερη, με περισσότερο ζήλο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν ε, στη φάση αλλαγής της έτσι κι αλλιώς. Το κοινοβούλιο είχε εκλογές. Η ανησυχία μας ήταν να μην γίνει υπαναχώρηση για αυτά τα βασικά ζητήματα. Ας πούμε αυτό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή της ε, επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό επιλέξαμε κάποια θέματα προτεραιότητας. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί στην ε, εισαγωγή νέων θεμάτων. Το θέμα της κοινή εκπαίδευσης λοιπόν των δικαστικών λειτουργών μας απασχόλησε και ως κληροδότημα της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Σεβόμενη πλήρως της αρμοδιότητας του Κοινοβουλίου, θεωρώ ότι η νέα φάση εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ορισμένα μόνο σημεία. Είναι πολύ σημαντικά όσα έχει κάνει η δική σας Επιτροπή ως τώρα, αλλά είναι και ευρύτατο το φάσμα που καλύψατε. Δεν είναι απλό να πάρει κανείς ε, αφορμή από όλα όσα έχουν γίνει και να τα μεταφράσει σε νέους κανόνες ο συσχετισμό μεταξύ οργανωμένου εγκλήματο και δημοσιονομικών οικονομία, δηλαδή η ροή κεφαλαίων. Αυτό είναι ένα καθοριστικό ζήτημα επί του οποίου καλό θα ήταν να υπάρξει όθηση στα πλαίσια τη Νέα Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Ιδίω και για τα περιουσιακά στοιχεία. Εδώ έγιναν κάποια βήματα πρόοδου, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ως προς Ως προς τους αλλοδαπούς μαθητές, να υπογραμμίσω κάτι περίεργο που χρειάστηκε να συζητήσουμε και παρουσία του συναδέλφου μου, του κυρίου Αλφάνου, Αλφάνου του Υπουργού Εσωτερικών, διότι από το έργο των Υπουργείων Εσωτερικών προέκυπτε ότι στις νομοθεσίες μας υπήρχαν κενά και να ως προς τον ειδικό χαρακτηρισμό των εγκλημάτων που σχετίζονται με τις παράλληλες συμπεριφορές, τις συμπεριφορές που οδηγούν σε τέτοιου είδου εγκληματικές ενέργειες. Το παραδέχτηκαν όλοι οι υπουργοί ενώ είναι διαφορετικό το επίπεδο προθυμίας να ορίσουμε καινούς κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είναι σημαντικό ότι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί το θέμα αυτό να είναι κοινή. Ακόμη και αν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στις εσωτερικές νομοθεσίες, στις κρατικές νομοθεσίες. Η νομική ορολογία είναι κάποιες φορές πολύ περιπλοκή. Δηλαδή, οι κανόνες εντοπίζουν κάποιες φορές συμπεριφορέ που είναι πολύ κοντά στην εγκληματική δράση αλλά δεν μπορούν να την ε, εντοπίσουν συγκεκριμένα. Λόγω χάρη κάποια ταξίδια, κάποιες μετακινήσεις. Το να προβλέψουμε τώρα πολύ με διαφορετικές ε, προδιαγραφές μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αποκλήσεις. Ας θυμηθούμε ότι έγινε το 70 και το 80 με την ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία στην Ήπειρό μα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντιφάσει μεταξύ των νομοθεσιών, διότι έτσι θα δώσουμε θύλακες όπου θα μπορέσουν, θα προσφέρουμε θύλακες όπου θα μπορέσουν να αναπτυχθούν τέτοιου είδου φαινόμενα εις βάρος των κρατών μελών. Ακόμη λοιπόν και δεν υπάρξει απόλυτη προθυμία, που δεν είναι δεδομένη, να έχουμε μια κοινή νομοθεσία, τουλάχιστον να υπάρξει προθυμία να έχουμε κοινή γλώσσα όταν περιγράφουμε το φαινόμενο αυτό. και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύνολο κοινών κανόνων σε ό,τι αφορά. Νομίζω ότι απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις, όλες τις βασικές ερωτήσεις για τα ντοσιέ που συζητήσαμε στη διάρκεια του εξαμήνου. Δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε να είμαστε πλήρως αισιόδοξοι, αλλά Παρά την τεράστια δουλειά που είχε γίνει από την ελληνική προεδρία και παρόλα που μπορούσαμε να βάλουμε το λέξη τέλος ε, την έκβαση κάποιων διαδικασιών, εμείς δώσαμε συνέχεια σε αυτά. Ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω ότι τουλάχιστον διατηρήσαμε την κατεύθυνση που έχει στόχο να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της, ε, του λειτουργήματος αυτού του οργανισμού αυτού. Το πρόβλημα που είχαμε συζητήσει στην τελευταία θητεία ήταν το θέμα της συλλογικότητας. Το κατά πόσον τα κράτη-μέλη δεν θα αλλάξουν τίποτα στις ποινικέ τους διαδικασίες ε, στην εσωτερική τους νομοθεσία, αλλά κάναμε μία πρόοδο διότι χώρε που ήταν πολύ εχθρικές ως προς τη δική μας κατεύθυνση, στο τελευταίο Συμβούλιο έδειξαν ε, διάθεση ανοίγματο προκειμένου να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της κεντρικής φυσιογνωμίας ε, αυτού του οικοδομήματος. Ακόμη όμως και αν τελειώνουν εδώ οι διαπραγματεύσεις, το γεγονός ότι εντοπίσαμε μια φυσιογνωμία, ε, μια, ένα σχηματισμό αυτόνομα από τα κάτι μέλη, ουσιαστικά διαφυλάσσει το λόγο ύπαρξη αυτού του οργανισμού, που δεν θα είναι μια απλή επανάληψη των εθνικών εισαγγελιών. Δεν θα έχει απλώς το ρόλο συντονισμού των εθνικών εισαγγελιών. Θα πρέπει να είναι ένα υποκείμενο που να λάβει ευρωπαϊκή ανάσα και ανεξαρτησία ω προ τα κράτη-μέλη αυτό το έμβριο, αυτό το ε, στοιχείο ε, σε εμβριακή κατάσταση, αν θέλετε, αυτός ο σπόρος για το μέλλον είναι ήδη πολύ σημαντικό. Είναι ένα βήμα πρόοδου που πρέπει να το διατηρήσουμε και χωρί υπερβολική ε, αισιοδοξία θεωρώ ότι κάναμε μια αποφασιστική κίνηση. Thank you. Ευχαριστούμε. Ήσασταν περιεκτικότατος ε, στις απαντήσεις σας. Μπορούμε να περάσουμε στο τμήμα εσωτερικές υποθέσεις με τον Υπουργό Αλφάνο. τον Υπουργό Εσωτερικών, καλώς ορίσατε. Και εσείς φυσικά θα μας παρουσιάσετε τον απολογισμό της Ιταλικής Προεδρίας στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Συμμετείχατε στην ε, Υπουργική Διάσκεψη G6 στο Παρίσι. Καλό θα ήταν να μας κάνετε και μια σύντομη αναφορά για αυτήν την Υπουργική Διάσκεψη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για την ευκαιρία που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε τα βασικά αποτελέσματα, τις βασικές εξελίξεις στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Από πολιτικής σκοπιάς πρέπει να πούμε ότι η Ιταλία ανέλαβε την Προεδρία αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ σε μια στιγμή ιδιαίτερα ευαίσθητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν διακυβευόταν η ίδια η Ένωση. Αλλά και για τις πολιτικές του χώρου εσωτερικών όπου οι ε, προθεσμίες, οι διορίες του προγράμματος της Στοκχόλμης αναθεωρήθηκαν από τις κατευθύνες γραμμές του Συμβουλίου τον περασμένο Ιούνιο. Η Ιταλία προσπάθησε να διατηρήσει τη συνέχεια με τις πρωτοβουλίες που είχαν ήδη αναλυφθεί στο παρελθόν βάσει των θεσμικών επιταγών, αλλά να συμπεριλάβει και τα, τις συνεισφορές των νέων κατευθυντήνων γραμμών για να αναπτυχθεί αντώνη δραστηριότητα που τώρα θα την παραδώσουμε στα χέρια των επόμενων προεδριών της Λετωνικής και της Λουξεμβουργιανής με τις οποίες μοιραζόμαστε το τρίο προεδριών. Τα θέματα της μετανάστευσης βρέθηκαν στο κέντρο των προτεραιοτήτων μας με το άτυπο συμβούλιο του Μιλάνου, όπου αντιμετωπίσαμε ρεαλιστικά το θέμα του τρόπου αντιμετώπισης της μεταναστευτικής πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πορεία που χάραξε η συζήτηση αυτή στο Μιλάνο, και το ίδιο στον απόϊχο της λειτουργίας της ομάδας δράσης για την Μεσόγειο, το Συμβούλιο του περασμένου Οκτωβρίου ε, ενέκρινε ένα κείμενο συμπερασμάτων με δράσεις για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δράσεις που πρέπει να αναλυθούν για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Η υλοποίηση των συμπερασμάτων αυτών μπορεί να είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση που ε, περιγράψαμε για έναν δραστηριότερο ρόλο και πιο αλληλέγγυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα λεπτομερές έγγραφο με κεντρικούς στόχους για ένα πρότυπο ε, διαρθρωμένης απόκρισης σε καταστάσεις πίεσης, ιδιαίτερο στη Μεσόγειο, ένα μοντέλο, ένα πρότυπο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, και αυτό δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να ε, αξιοποιηθεί και σε άλλους γεωγραφικούς όρους, διότι όχι μόνο η Μεσόγειος προκαλεί ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εκκίνηση μιας νέας φάσης στην φύλαξη των μεσογειακών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στην επιχείρηση τρίτονας της ε, Frontex. Πρόκειται για ένα μεγάλο αποτέλεσμα, όχι μόνο για την Ιταλική Προεδρία που ε, έκανε σοβαρές προσπάθειες γι' αυτό, αλλά και του έργου της ε, Ομάδας Κρούσης για την Μεσόγειο και ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτέλου δίνει ένα ηχηρό μήνυμα για τον έλεγχο των εξωτερικών της συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πέρα της συνδυασμένης φύλαξης των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμπεράσματα επικεντρώθηκαν και στη βελτίωση του συστήματος υποδοχής και συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Κάτι που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη αξία για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της μετανάστευσης. Η μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ούτως ή άλλως ένα δεδομένο που είναι δομικό. Ένα δεδομένο δομικό το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ερχόμενα χρόνια. Υπ' αυτού ε, αυτή τη άποψη είναι σημαντικό να υπάρξει ενίσχυση της ευρωπαϊκή δράσης και σε τρίτες χώρες και με σκοπό να ελέγξουμε τις επανειλημμένες, ε, ε, την, επανα, ε, την επανειλημμένη και την εντατική αναχώρηση μεταναστών αλλά το ίδιο και την εμπορία ανθρώπων ώστε να αντιμετωπιστεί η λαθρομετανάστευση. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν προσέγγιση, συνολική προσέγγιση για τη μετανάστευση από το 2005 ε, έχει ήδη ενισχυθεί και δίνουμε έμφαση σε εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας που έχουν εγκριθεί αλλά και ενδεχόμενε μελλοντικέ νέε συμφωνίε με τρίτε χώρε όπω αυτή με την Ιγυρία που πρόκειται να υπογραφεί. Είναι σαφέ ότι τα διάφορα πολιτικά σκηνικά των διαφόρων χωρών μα φέρνουν αντιμέτωπου με εμπόδια πολύ σοβαρά για την κίνηση δράσεων συνεργασία όπω συμβαίνει με τη Λιβύη. Όμω, αλλού χρειάζεται και μεγαλύτερη πυγμή για να υποχρεώσουμε τι χώρε που είναι έτοιμε να συνεργαστούν να το κάνουν. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε την ε, ε, συνεργασία με, τις πολυ... με τους πολυμερείς ε, διεθνείς οργανισμούς που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα την τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους, για τους πρόσφυγες, καθώς και το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση. Για να ενισχυθούν αυτές οι προσπάθειες πρέπει να υπάρξουν θετικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών του τομέα των ιστορικών υποθέσεων και της εξωτερικής ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε κοινή στόχη και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα να τα αποσπάσουμε σύντομα. Είπα αυτό το οπτικό πρίσμα η Ιταλική Προεδρία στα τελευταία συμβούλια εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης φρόντισε να υπάρξει συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και οργάνωσε στη Ρώμη στις 27 Νοεμβρίου του 2014 μια σημαντική διάσκεψη, κοινή διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι η πορεία αυτή που έτυχε ευρεία στήριξη θα συνεχιστεί για πρώτη φορά διαρθρωτικά οργανώθηκε ένας γύρος συζήτησης με υπουργούς εσωτερικών και εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 Νοεμβρίου στη Ρώμη ως ε, μετάφραση του ατύπου των συμπερασμάτων μιας σύστασης του Ατύπου Συμβουλίου του Μιλάνου του περασμένου Ιουνίου. Έπειτα, στις 28 Νοεμβρίου στη Ρώμη οργανώθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων της διαδικασίας του Ραμπάτ. Μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου με τους, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκπροσώπων των χωρών της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής με σκοπό την ανάπτυξη επίσης στη Ρώμη. Οργανώθηκε η συνάντησή με τους εκπροσώπους των χωρών του κέρατος της Αφρικής, ώστε να έχουμε έναν πιο διαρθρωμένο διάλογο για τα θέματα της μετανάστευσης και μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδικασίας του Ραμπάτ, ώστε να ε, εφαρμοστεί ενδεχομένω και σε άλλες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα των διεθνών αυτών ε, εξελίξεων μας ανησυχούν ακόμη, διότι η αστάθεια στη Λιβύη που κατευθείαν οδήγησε μεταναστευτικέ ζωέ προ την Ιταλία είναι ένα ε, πραγματικά ε, ξεχωριστό παράδειγμα, αλλά όχι απομονωμένο. Η πίεση και η ροή ε, προσφύγων που έρχονται από τη Συρία μπορεί να πάρει δραματικές διαστάσεις και να αποσταθεροποιήσει τις γειτονικέ όμορες χώρες με τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες πιο καταστροφικές από τις σημερινές. Το θέμα των ετούντων άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη εκπροσωπεί λοιπόν μια πρόκληση εντός της πρόκλησης. Μια πρόκληση εν την προκλήση. Και αυτό προκειμένου να υπάρξει μια σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Πέρυσι εγκρίθηκε μια σειρά από κανόνε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση που επέτρεψε να συμπληρωθεί η δεύτερη φάση της, του λεγόμενου κοινού συστήμα, Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Η Ιταλική κυβέρνηση, όπως και οι κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών, δεσμεύτηκε να υλοποιήσει το σύστημα αυτό σε συμφωνία με τους στόχους που ορίζουν οι νέες στατικικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα των εσωτερικών, όπως εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26-27 Ιουνίου 2014. Πρόκειται για έναν σημαντικό στόχο στον δρόμο που θα μας οδηγήσει σε διαδικασίες και επίπεδα υποδοχής ομοιογενέστερα μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, είναι πεποίθησή μου ότι απαιτούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον βήματα πρόοδου. Ιδιαιτέρως πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά προς έναν μηχανισμό αμοιβές αναγνώρισης των αποφάσεων σε θέματα ασύλου και προς αυτό το σκοπό η Ιταλική Προεδρία ξεκίνησε την μελέτη σε τεχνικό επίπεδο γνωρίζοντας ότι αυτός ο στόχος βεβαίως είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον έχουμε ε, την εμπιστοσύνη ότι οι άοκνες προσπάθειες της Ιταλικής Προεδρίας για να τροποποιηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου σε ό,τι αφορά τους κανόνες των ασυνόδευτων ανηλίκων, πρόταση που έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο, μπορεί να τύχουν ευνοϊκής προώθησης από την Λεπτονική Προεδρία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ε, διαρθρωμένη συζήτηση μεταξύ των ομελών με ε, σχέδια για την δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες διέλευσης και που θα ε, δημιουργηθούν επιτόπου σε συνεργασία με την υπατερμοστία του ΟΗΕ στην ε, διαδικασία εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Έτσι θα υπάρξει ανακατανομή της άφηξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια οπτική γωνία αλληλεγγύης ανάλογα με την ε, θελούσια δράση των κατών μελών. Επίσης, τα θεμελιώδη εργαλεία για την ε, καλλιέργεια της ε, νόμιμης μετανάστευσης και την δημιουργία σχέσεων καλής πίστης με τις τρίτες χώρες θα μας βοηθήσει και με το πακέτο μέτρων FEE e, σύνορα, Smart Borders. Θέλουμε καλέ σχέσει με τι τρίτε χώρε και του πολίτε του για να ε, αυξηθούν και οι πρόπτυχε ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των χωρών προέλευση των μεταναστών. Είπα αυτήν, προς αυτήν την ε, κατεύθυνση ε, Αντίναμε τις προσπάθειες διαπραγματεύσεων για την πρόταση οδηγίας για τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής των πολιτών των τρίτων χωρών για σκοπούς έρευνας και σπουδών και ελπίζουμε ότι στο δυνατόν συντομότερα θα μπορέσει να ξεκινήσει και η όλη συζήτηση με το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, η Προεδρία έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ρίζος, ρίζ, της ριζοσπαστικοποίησης, τη τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και όλων των εγκληματικών φαινομένων που έχουν να κάνουν με τη λαθρομετανάστευση όπως την εμπορία ε, και την ε, πώληση ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά το κυβερνοέγκλημα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και η νέα στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκή Ένωση, του χρόνου. Η Ιταλική Προεδρία και επειδή στην προετοιμασία αυτού του σημαντικού εγγράφου ξεκίνησε με το κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της 5 η Δεκεμβρίου 2014. Πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη μνήμα και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό η Ιταλία πρότεινε και πέτυχε την έγκριση από την πλευρά του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της περασμένης 5ης Δεκεμβρίου 2014 ένα κείμενο συμπερασμάτων για την καταπολέμηση της διείσδυσης μελών οργανωμένου ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην νόμιμη οικονομία μέσω της ανείχνευσης και την παρακολούθηση των δημοσιονομικών ροών, ιδίως στους δημόσιους διαγωνισμούς. Είναι πολύ περίπλοκη η διοργάνωση και οι διεθνείς προεκτάσεις του οργανωμένου εγκλήματος, γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη επίγνωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης του όλου θέματος και ανάληψη ευθυνών ώστε οι, αρχές, οι αρχές των κρατών να λάβουν δράση. Υπ' αυτήν την οπτική γωνία προωθήσαμε και τη δημιουργία ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού δικτύου για την αντιμετώπιση οργανωμένων ε, ομάδων οργανωμένου εγκλήματος με χαρακτηριστικά μαφίας κάτι που εγκρίθηκε και από το, ε, από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στις 5 Δεκεμβρίου 2014. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η Ιταλική Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο φαινόμενο των foreign fighters, των αλλοδαπών μαχητών μετά το Συμβούλιο 30 Αυγούστου 2014 και επειδή μας ζητήθηκε να επιταχύνουμε και να εμβαθύνουμε τα μέτρα που σκοπό έχουν να εμποδίσουν την ε, μετακίνηση μαχητών προς το Ιράκ και τη Συρία, η Ιταλική Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη προτεραιότητα στο θέμα. Το Συμβούλιο Τζάι συζήτησε το θέμα στις συνεδριάσεις του, του, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου θύμισε ότι πρέπει να ε, αναλυθούν κάποια ειδικά μέτρα με κατεπίγουσα ταχύτητα και οι υπουργοί ε, πρότειναν την ένταση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων χωρίς διακριτικές μεταχειρήσεις. Αυτό μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μεσοπρόθεσμα πρέπει να αναζητηθούν οι κατάλληλε βελτιώσει ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για του αλλοδαπού μαχητέ. Πολλά συστήματα, δυνατά συστήματα συζητήθηκαν του περασμένου μήνε, ιδίω ω προ το ΣΥΣ 2 και τα αναλυτικά ντοσιέ τη Europol. Επίση, το Συμβούλιο εξέτασε το πώς μπορεί να ε, βελτιώσει την νομική αντιμετώπιση του θέματος για να αντιμετωπίσουμε την στρατολόγηση και την ριζοσπαστικοποίηση, το Συμβούλιο ανέκρινε μια σειρά από κατευθυντήριε γραμμέ. Κατευθυντήριε γραμμέ τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση και την στρατολόγηση. Αυτό είναι ο ορισμό. Αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ έχουν ιδιαίτερη σημασία ω προ το φαινόμενο των αλλοδαπών μαχητών και σκοπό έχουν να δημιουργήσουν μια στρατηγική αντιριζοσπαστικοποίησης όπως εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2014. Οι ε, συγκεκριμένες δράσεις που προβλέπει από τις συντεκτήρε γραμμές έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται από τα ενδιαφερόμενα Για να αναχαιτήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση στον κυβερνοχώρο, στις 8 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, πριν από το Συμβούλιο Τζάι, οργανώσαμε ένα άτυπο δείπνο, μια άτυπη συνάντηση με τις τεράστιες εταιρείες του διαδικτύου, με τους κολοσσούς του διαδικτύου, θεωρώντας ότι οι εταιρείες αυτές εκπροσωπούν την χρονική συγκυρία όπου έρχονται σε επαφή και οργανώνονται διάφορες κοινότητες. Οπότε η επίθεση μετά δεν γίνεται κατά των κυβερνήσεων αλλά κατά των λαών. Πρέπει να βρούμε λοιπόν νέες μορφές συνεργασίας για τα δικαιώματα σε συνεργασία με τις ε, ε, μεγαλύτερες εταιρείες του διαδικτύου. Η Ιταλική Προεδρία έδωσε μεγάλη σημασία και στην υλοποίηση των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας εντός των διαφόρων τεχνικών ομάδων εργασίας. Έτσι μπορέσαμε να έχουμε μια σημαντική βελτίωση της όλης πορείας. Ταυτόχρονα να επισημάνω ότι όλη η απειλή είναι πολύ σοβαρή και πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Το Συμβούλιο Τζάι σε συνεργασία με το συντονιστή για τα θέματα τρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσει όλες τις ανάλογες δράσεις. Επίσης, την διάρκεια του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου έγινε και μία ενδελεχής συζήτηση για το θέμα των αλλοδαπών μαχητών ιδίως σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και δύο συγκεκριμένε τους πτυχές ή απέτηση να ξεκινήσει, να συνεχιστεί η όλη διαδικασία και η συζήτηση για το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τον κατάλογο επιβατών, αλλά και την ένταση φύλαξης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων με πλήρη αξιοποίηση του συστήματος SIS-2. Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε με μια σειρά από συγκεκριμένε δράσεις. Ενέκρινε 22 μέτρα από τον Ιούνιο που είχαν ήδη προταθεί από τον Ιούνιο 2013 και από τον συντονιστή για την καταπολέμηση της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει δική μας πρότασης, ταλικής πρότασης, προτάθηκε να αξιοποιηθεί και η ιδέα των πολυεθνικών ad hoc ομάδων για το φαινόμενο των αλλοδαπών μαχητών και προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και στο λειτουργικό επίπεδο, το επιχειρησιακό επίπεδο για την καταπολέμηση των αλλοδαπών μαχητών. Η Ιταλική Προεδρία ξεκίνησε και σχεδίασε ένα εγχείρημα, ένα μια άσκηση σε συνεργασία με τη Europol για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με σημεία επαφή κατά τη τρομοκρατία, ιδίω για την περίπτωση των αλλοδαπών μαχητών. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει και ένα λειτουργικό πρωτόκολλο για να λειτουργήσει αυτό στα περισσότερα κράτη-μέλη. Επίση, με αφορμή το πρόσφατο συμβούλιο Τζάι, κατατίστηκαν μια σειρά από κατευθυντήριε γραμμέ για την υλοποίηση τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση από τρομοκρατικέ ομάδε. Ωραία. Ολοκληρώνοντας αυτή την παρέμβαση, ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να έχουμε εδώ διάλογο που δείχνει πόσο επικοδομητική είναι η επαφή μεταξύ των θεσμικών οργάνων και είμαι πεπισμένος ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ε, μια μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου με μοναδικό στόχο, παρόλο που οι θέσεις κάποιες φορές διαφέρουν, με μοναδικό στόχο να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη ελευθερότερη και ασφαλέστερη. Ευχαριστώ. Ε, mm, Πρόεδρε, να προσθέσω ότι στη σύνοδο G6 στο Παρίσι δεν απήντησα στη συγκεκριμένη σας ερώτηση, διότι πρόκειται για μία διάσκεψη άτυπη, με καμία δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Αυτό οργανώθηκε υπό Γαλλικής Προεδρίας στι 6 Νοεμβρίου στο Παρίσι, οπότε ο συνάδελφος Κάσινευ θα μπορούσε να μας πει τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να ε, υπερχιλήσω τις παρεμβάσεις μου σε έναν τομέα που δεν είναι ο Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιεκτικότατη παρουσίαση των συμπερασμάτων σας. Εννέα ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο, είναι αρκετή και ο χρόνος λίγος. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι και να περιοριστείτε στα δύο λεπτά το πολύ ο καθένας. Επίσης, παρακαλώ να μην μιλάτε πολύ γρήγορα, έτσι ώστε οι διερμηνείς να μπορέσουν να μεταφράσουν αυτά που λέτε. Κυρία Μετσόλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε εκτενέστατα τον απολογισμό σας. Θα ήθελα να εστιάσω σε κάποια σημεία και μετά οι συνάδελφοι θα κάνουν τις δικές τους, τους ερωτήσεις. Μετανάστευση. Όπως είπατε, η Ιταλία έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, διάσωση σε επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο μέσω του προγράμματος Mare Nostrum, το οποίο ήταν ένα μόνο μερές πρόγραμμα, το οποίο επίσης έφτασε στο τέλος του. Μετά τα γεγονότα στη Λαμπεντούσα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα πάρα πολύ σημαντικό ψήφισμα, στο οποίο υπήρχε συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων και αναφερόταν η συνέχεια στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Στο ψήφισμα αυτό είχαμε ζητήσει την ε, δημιουργία ενός ε, μηχανισμού βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος θα μείωνε την πίεση που δέχονταν ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία δέχονται το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου και ετοιμάτων προστασίας. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι πρόοδος έχει γίνει από το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Επίσης, όσον αφορά την επαναγκατάσταση, είναι κάτι που αφορά τη χώρα μου τη Μάλτα πάρα πολύ. Θα ήθελα να μάθω περισσότερες πληροφορίες. Έχουν γίνει αλλαγές σχετικά με τις υποσχέσεις δεσμεύσεις κρατών μαλλιών να βοηθήσουν άλλα κρατημέλη. Γνωρίζω πως έχουν γίνει πριν από κάποια χρόνια κάποιες αλλαγές, όμως έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει κάτι από τότε. Έπειτα, είστε ικανοποιημένος με την απάντηση της Frontex όταν άρχισε η επιχείρηση τρίτονας. Θεωρείτε πώς θα είναι επιτυχή σε σχέση με την επιτυχία του προγράμματος Nostrum; Διότι νομίζω πως συμφωνούμε όλοι για το ότι η επιχείρηση τρίτων θα είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση μόνο εάν έχουν τα κράτη-μέλη τους κατάλληλους πόρους και δεδομένη τη κατάσταση με του πόρου, θα μπορούσατε εσεί να μα ενημερώσετε για το αν έχει γίνει κάποια πρόοδο σχετικά με την ε, διάθεση των πόρων αυτών από τα κράτη-μέλη. Τέλο, στρατηγική ασφαλεία. Αυτή τη στιγμή συζητούνται οι προτεραιότητες. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης της αύξησης του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης. Ελπίζω να μου απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μετσόλα. Η κυρία Τσινίτσι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, κύριε Υπουργέ για την πλήρη παρουσίασή σας για το έργο αυτό που συμπλήρωσε και την παρουσίαση του κυρίου Ουρλάντο. Πολλά έγιναν στη διάρκεια του Ιταλικού εξαμήνου. για να έχουμε νέους κανόνες στον ιστορικό χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τέλος πάντων τέθηκαν τα θεμέλια για μια μεγαλύτερη ενοποίηση από την ερχόμενη Προεδρία που θα πρέπει να δουλέψει σε θέματα που αναφέρατε. Ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές διότι εργάστηκα πολλά χρόνια για τα θέματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Στην παρουσίασή σας κάνατε λόγο για τους αλλοδαπούς ασυνόδευτους ανηλίκους. Και επειδή ο Πρόεδρος δεν μας έχει δώσει πολύ χρόνο, πολύ συνοπτικά να ρωτήσω. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περιττέρω για τις συγκεκριμένες ε, δράσεις που προβλέφθηκαν, για μέτρα που μελετώνται για τους αλλοδαπού ασυνόδευτου ανήλικου που είναι πολύ άρεθμοι στην επικρατειά μας αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι υπολογισμοί και αριθμητικά στοιχεία και ω προ την υποδοχή και ω προ τι αιτήσει ασύλου. Και μπορείτε να μας πείτε και κάτι παραπάνω για τις δράσεις αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος που ακριβώς ασχολείται με την εμπορία τη διακίνηση ανθρώπων, διότι πολλές φορές ακριβώς αυτοί οι αλλοδαποί ασυνόδευτοι ανήλικοι πέφτουν στα χέρια των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και ε, είναι και αντικείμενα ε, σοβαρού εγκλήματος διακριτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ακόμα ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο και για να μπορέσω να δώσω τη δυνατότητα στους υπουργού να απαντήσουν, δυστυχώς πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Κάρλος Κοέλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Νότας. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τελική Προεδρία για τη δουλειά που έκανε. Ήταν υποδειγματική η συνεργασία που είχατε με το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσω διότι αποδώσατε ιδιαίτερη σημασία στις μεταναστευτικές ροές και την κατάσταση στη Μεσόγειο. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μια οριστική προσέγγιση για τη Μεσόγειο και για τις μεταναστευτικές δροές. Ταυτόχρονα όμως βραχυπρόθεσμα πρέπει να δράσουμε για να αποφύγουμε να γίνει το κημητήριο της Ευρώπης ε, η Μεσόγειος, ε, όπως είδαμε με τις τελευταίες εξελίξεις και το συζητήσαμε στο Στρασβούργο. Ήθελα να πω μόνο πως ε, απογοητεύτηκα με τη θέση που έλεγε το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου για την αξιολόγηση του Σέγγεν. Εγώ περίμενα το Συμβούλιο να διευκολύνει τη θέση σε ισχύ του νέου μοντέλου λειτουργίας και να ε, δηλώσει απερίφραστα την υποστήριξή του για τα νέα εργαλεία που θα υποστηρίξουν το σύστημα αξιολόγησης. Όμως δεν έκανε αυτό ε, το Συμβούλιο. Ε, δεν λειτουργήσε η αξιολόγηση τα τελευταία 15 χρόνια. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ε, δημιουργήθηκαν δύο μέτρα και δύο σταθμά. υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης για τις χώρες που ήθελαν να μπουν στο χώρο Σέγγεν, Βουλγαρία, Ρουμανία. Ε, όμως ε, δεν εφαρμόστηκαν τέτοια κριτήρια για όσους ήταν ήδη στο χώρο Σέγγεν. Και φαίνεται ότι το Συμβούλιο θέλει να επιστρέψει στο παρελθόν όπου ε, ήταν διακυβερνητικό εργαλείο και όχι ευρωπαϊκό ε, το σύστημα, ο χώρος Σέγγεν. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκανε το Συμβούλιο. Uh, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σλέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Υπουργό για την εισήγηση. Ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα σε σχέση με την επιχείρηση Τρίτονα. Είπατε ότι είστε θετικός και ότι πάει προς τη σωστή κατεύθυνση δημιουργίες κοινών ευθυνών για μια πρόκληση που δεν μπορεί να είναι μόνον ευθύνη των συνοριακών χωρών της Επίρου. Πρέπει να θεωρηθεί ευρωπαϊκό πρόβλημα. Όμως έχουν εγερθεί πολλά ερωτηματικά. Δεν το η επιχείρηση τρίτονας. Δεν έχει τη διαθέση της τα ίδια μέσα. Είναι πολύ χειρότερα μάλιστα σε σχέση με αυτό που είχε προβλέψει η Ιταλική κυβέρνηση με τον Μάρε Νόστρουμ. Όμως υπάρχει και θέμα τομέων παρέμβαση, παρέμβασης με 72 μίλια ή 30 από τις Ιταλικές ακτές και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι τη αποτελεσματική επιχείρηση τρίτονα με όσο ήταν η Μαρενόστρουμ. Επίση υπάρχει ανησυχητική παρατήρηση του ε, πρόεδρου τη Frontex. Τι μπορείτε να μα πείτε λοιπόν ω προ τον απολογισμό των δράσεων αυτό το πρώτο μήνα λειτουργία. Να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το πρόβλημα θα λυθεί μειώνοντας τον τομέα παρέμβασής μας. Εγώ έχω την αντίποση ότι αντιθέτως θα έχουμε καινούργια ναυάγια και απλώς δεν θα βλέπουμε όσους ε, έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Μια θάλασσα που έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό ε, νεκροταφείο με κάτω από τον ουρανό, ενώ το πραγματικό νεκροταφείο δεν έχουμε κοινή πολιτική ασύλου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Μόλις ένα πράγμα προλαβαίνω να σας ρωτήσω, αλλά ήδη το έθιξε η συνάδελφος για το Μαρενόστρουμ και το συσχετισμό με την επιχείρηση Τρίτονας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιος δεν μας λέει την αλήθεια. Εσείς λέτε ότι η Ευρώπη ανέλαβε με τη Frontex αρμοδιότητες που δεν μπορούσε πλέον να επομίζεται μόνη της Ιταλία. Επιπλέον λέτε ότι ο Κλάους Ρόσλερ ε, στην ε, Προεδρία της Frontex δηλώνει ότι είναι πάρα πολλές οι αποστολές διάσωσης της Ιταλίας εκτός του τομέα της, το 30 ναυτικά μίλια που ορίζει η Ένωση. Η επιχείρηση, λέει πάλι ο πρόεδρος της Frontex, δεν συνάδει με το επιχειρησιακό πρόγραμμα και δεν θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Ποιος λέει ψέματα σε ποιον σε αυτή τη θλιβερή ιστορία, κύριε Υπουργέ. Σας ερωτώ σε αυτό το τέλος ε, εξαμήνου, δεν χρειάζονται σοβαρές διευκρινήσεις από τη Frontex. Δεν πρέπει να καλέσετε τον οργανισμό να σεβαστεί τους κανόνες που ορίστηκαν στο τέλος του 2013. Την υποχρεώνουν όχι μόνο να προστατεύει τα σύνορα, αλλά να προχωρεί και σε ενέργειες έρευνας και διάσωσης και να εφαρμόζει και το δίκαιο της θάλασσας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα Υπουργέ Αλφάνου. Και εγώ να επανέλθω στην επιχείρηση τρίτονας όπως είπαν οι συνάδελφοι Σχάιν και Σπινέλη. Ήθελα περισσότερα στοιχεία για αυτή την επιχείρηση. Είπατε προηγουμένως ότι μιλάμε για έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, αλλά στη διάρκεια συνεδρίου που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συνοβούλιο στην Κατάνια τον περασμένο μήνα υπήρχαν εκπρόσωποι της Ιταλική, του Ιταλικού Ναυτικού που, της Ιταλικής Ακτοφυλακής μάλλον που είπαν ότι η επιχείρηση έχει, παρα, έχει με προχωρήσει και σε ε, ενέργειες διάσωσης, έρευνας και διάσωσης πέραν της προστασίας των εξωτερικών ε, σύνορων. Και επαναλαμβάνω, πέραν των 30 ναυτικών μιλίων μπορεί να υπάρξουν ενέργειες ε, έρευνας και διάσωσης. Εκεί θέλαμε διευκρίνηση. Όπως διευκρίνηση χρειάζεται και η διαδικασία του χατούμ. Είπατε προηγουμένως στην εισηγήσή σας κάποια πράγματα και Λέτε ότι χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με σχέδια συνεργασία, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, με τη συνεργασία των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τη μετανάστευση και με την υπατιαρμοστία του ΟΗΕ. Όμως, επί τη ουσία δεν είναι σαφέ τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα σχέδια, ποιος θα συμμετέχει. Πολλοί είναι ε, ε, αυτοί που εκφράζουν ε, μη ικανοποίηση και φόβους για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι γίνεται λοιπόν με τη διαδικασία του Χαρτούμ που και αυτό, αυτή ξεκίνησε τον περασμένο μήνα και είπατε ότι στη διάρκεια του Ιταλικού εξαμένου τη Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων συζητήθηκε και η βελτίωση των συστημάτων υποδοχή. Να πω ότι θεωρώ πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση των χώρων υποδοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε το δικό μα παράδειγμα τη Ιταλία για τα πρόσφατα σκάνδαλα σε σχέση με τι παρισπρήσει των μελών τη μαφία σε κέντρα υποδοχής το ίδιο και η Ελλάδα. Ε, εδώ λοιπόν τι μπορείτε να πείτε για την ανείχνευση των ε, ε, μεταναστευτικών ροών και πώς θα αναλυφθεί η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των δράσεων της μαθής και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει πάντοτε να αγωνιζόμαστε και να είμαστε σε επαγρύπνηση για το πώς οι οργανωμένες ομάδες και με χαρακτηριστικά μαφία, μπορεί να εκμεταλλεύονται την απελπισία των ετούντων άσυλο. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, έχουμε ακόμη πολλούς ε, που έχουν εγγραφεί. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ να παραμένετε στο ένα λεπτό ιδάλως. Ο χρόνος για τους υπουργού δεν θα φτάσει για να απαντήσουν σε όλα αυτά. Προσπαθείτε να περιοριστείτε σε ένα σημείο, σε ένα λεπτό. Κυρία Μπιόρκα, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομη. Η QNGL θεωρεί ότι η μεταναστευτική πολιτική ε, ξεκινάει από ένα σε εφαλτήριο, διότι ξεκινάμε από νομικά μέτρα αντί να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υποδοχή αυτών των ανθρώπων εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες, όμως ε, θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα βιώσιμο, ένα αξιοπρεπή τρόπο ε, και σύστημα υποδοχής αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν όταν διατυπώνουμε την πολιτική μας λαμβάνετε αυτό δεόντως υπόψη. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο ζητήματα και να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, προσπαθήσαμε ήδη, έχουμε κάνει μια ερώτηση για να μάθουμε ποια είναι τα αποτελέσματα, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Λοιπόν, ξανακάνω την ερώτηση. Ε, στο στην αποστολή πόσους ε, συλλάβατε και τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Ε, κρατούνται ακόμη κάπου σε κάποιο κέντρο ή έχουν επαναπροωθηθεί. Θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις στα νούμερα. Δεύτερον, η διαδικασία χαρτούμ. νουμερο νουμερα δευτερον ιδιαίτερα επικριτική ε, στάση σε σχέση με την εξωτερικοποίηση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται να συνεργαζόμαστε υπό αίρεση με τις ε, τρίτες χώρες, ε, δηλαδή υπό την αίρεση ότι θα ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές. Ε, δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε με την Ερυθρέα και το Σουδάν. Είναι δικτατορίες εκεί. Θέλουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα σταματήσω εδώ γιατί αλλιώς θα, δεν θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας Ευχαριστώ. Weinberg. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αλφάνου για την παρουσίαση που μας έκανε θα ήθελα να κάνω κάποιες διαπιστώσεις και κάποιες ερωτήσεις. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τους διακινητές και το λαθρεμπόριο ανθρώπων. Μεγενθύνεται διαρκώς το πρόβλημα. Πώς όμως πρέπει να ρυθμιστεί η κατάσταση, πώς θα σταματήσει αυτό το, το φαινόμενο ε, και αυτό πώς θα γίνει στα εσωτερικά αλλά και στα εσωτερικά σύνορα. Ε, μιλήσαμε επίσης για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε την οδηγία ε, για την μπλε κάρτα, τους εποχιακούς εργαζομένους ε, και μας είπατε ότι πρέπει να γίνεται screening, έλεγχος, ε, ώστε επιτόπου να κρίνουμε τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα υποχρεωθούν, αυτό εννοείται, να υποδέχονται τους μετανάστες ή κρίνεται ότι πρέπει να γίνει ένας επιμερισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα εφαρμόσετε την αλληλεγγύη ακριβώς, πώς θα έχετε έχετε ε, επιστρέφοντας ε, στην Σουηδία, μπορώ να σας πω ότι έχουμε 25 φορές με περισσότερους μετανάστες σε σχέση με την Ιταλία ετησίως. Ε, και Ε, θα πρέπει να υπάρχει επιτόπου ε, ε, υποδοχή στους πρόσφυγες, όπως είδαμε με την περίπτωση της Ιορδανής την περασμένη εβδομάδα. Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα της παροχής βοήθειας επιτόπου. Ευχαριστούμε, ο κύριος Γκεμπέγκ. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση του κύριου Ορλάντο στη δική μου ερώτηση ήταν πολύ σύντομη και όχι αρκετά ικανοποιητική. Ξανά λοιπόν θα ρωτήσω η οδηγία για την ίση μεταχείριση των εφηλεκισμένων ανεξάρτητα από ε, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό κτλ. Η οδηγία λοιπόν για την ίση μεταχείριση υπάρχει και είναι σε ισχύ. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που ανησυχούν ε, για το ότι η πρόταση αυτή, η οδηγία, αν εγκριθεί, θα περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Επίσης, εμένα με ανησυχία σάφια στη διατύπωση της οδηγίας αυτής, που θα έχει ενδεχομένως ε, ανεπιθύμητες ερμηνείες από τα κράτη-μέλη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πάνω από 100, 100 μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν υπογράψει μια επιστολή προς τον πρόεδρο Γιούνκερ και του έχουν ζητήσει να αποσύρει την ε, οδηγία αυτή. Σχετικά με αυτή την επιστολή θα ήθελα να ρωτήσω εσείς τι θα συμβουλεύατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ερχόμενη Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Κύριε Φοντάνα, έχει το λόγο τώρα. Ο κύριος Φοντάνα, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, ακόμα δεν έγινα εμεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Πολύ γρήγορα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι εάν υπάρχει σοβαρή διαφορά μεταξύ των όσων θα κάνει, των όσων κάνει η επιχείρηση τρίτων σε σχέση με το Μαρενόστρουμ. Διότι άκουσα πολλοί συνάδελφοι να λένε ότι το Mare Nostrum ήταν μια επιχείρηση διασωστική. Ναι, αλλά δυστυχώς και με την επιχείρηση αυτή υπήρξαν και πάρα πολύ μικροί από τους 12.000 ε, μετανάστες ε, που περιμέναμε 3.000 εξαφανίστηκαν στη θάλασσα. Ε, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Επίσης με τη σεξουαλική εκμετάλλευση τι γίνεται κύριε Υπουργέ σε σχέση με αυτό και νομίζω ότι και τα ταξίδια αυτά απελπισίας που καταλήγουν σε τραγωδίες ξέρουμε ότι έχουν συμβεί πολλά τέτοια επεισόδια και φέτος Δεν πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια στις χώρες προέλευσης των ανθρώπων αυτών όπου υπάρχουν ένοπλες σειράξεις, εκεί να αποφεύγεται η μετανάστευση, δηλαδή να μένουν οι άνθρωποι αυτοί στα σπίτια τους. Ξέρουμε ότι το 80% των ανθρώπων αυτών που φτάνουν στην επικράτειά μας έρχονται από τη Λιβύη. Όμως στην Ευρώπη κάποιο ε, είναι και κάπως υπεύθυνη για όσα συνέβησαν στη Λιβύη. Αφού η Ευρώπη λοιπόν σε μερικές περιοχές του κόσμου όπως τη Λιβύη και σε μέρη της Συρίας έχει επιφέρει κάποια προβλήματα και κάποιες ζημιές, ας αναλάβει και τις ευθύνες της. Ε, και σε ό,τι αφορά τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών Κάποιοι είναι λαθρομετανάστες εφόσον δεν τους εγκριθεί το άσυλο. Μπορεί να γίνει κάτι και για αυτούς. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντάλη. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Um... Υπόσχομαι, θα είμαι σύντομη. Κύριε Αλφάνο, για την ε, νόμιμη μετανάστευση, μιλήσατε για τις ε, νόμιμες μεταναστευτικές οδούς, κάτι με το οποίο ασχολείται επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα όμως να ε, να πω ότι υπάρχει διαφορά στις ε, αληθινές τάσεις των ε, διάφορων κρατών μέλων. Χρειαζόμαστε μια συνολική ολοκληρωμένη προσέγγιση και για το θέμα των νόμων μεταναστευτικών οδών. Στο έγγραφο που λάβαμε βλέπουμε την ανάγκη ενίσχυσης της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως παρατηρούμε κάποια κράτη-μέλη που έχουν τονίσει τη σημασία αυτής της πανεγκατάστασης και κάποια άλλα που θεωρούν ότι η επανεγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται μόνο με προαιρετική προσέγγιση. Αυτό δεν μου φαίνεται ε, πώς αντανακλά ε, την ευρωπαϊκή δέσμευση, ούτε πως δίνει μία λύση στην κατάσταση. Εσείς ποιες λύσεις προτείνετε ή ποιες εξετάζετε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση από εμένα. Αναφέρατε την συλλογή των ε, δεδομένων των επιβατών προσωπικών δεδομένων των επιβατών. Η γενική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μια πρόταση του 2012. Φέτος τον Απρίλιο είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, χρήση και κράτηση προσωπικών ε, δεδομένων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη του την απόφαση αυτή του δικαστηρίου και αν έχει αναθεωρήσει την άποψή του για ε, νομικά και πολιτικά για την πρακτική αυτή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Τώρα θα ήθελα εφόσον ακούσατε όλες τις ερωτήσεις, να απαντήσετε σε αυτές. Έχουμε 10 λεπτά και ενδεχομένως οι διεμηνείς να μπορέσουν να παραμείνουν λίγα λεπτά ακόμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε δέκα λεπτά, γιατί είναι πολύ άριθμα τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Ένα. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί πιο πολύ από όλα είναι η μετανάστευση. Δεν υπάρχει δράση που μπορεί μόνη της να αναχαιτήσει ένα φαινόμενο όπως αυτό της εμπορίας των ανθρώπων ή των ε, παράτυπων και παράνομων μεταναστεύσεων. Υπάρχει μία vision, μία κοινή θεώρηση και μια στρατηγική και εκεί θα πρέπει να εντοπίσουμε τις προσπάθειες όλων. Η στρατηγική προβλέπει δράσεις συνεργασίας με τις τρίτες χώρες της Μεσογείου και δράση της Frontex, Frontex στα θαλάσσια σύνορα, καθώς και ευρωπαϊκή δράση όπου θα πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα κοινό σύστημα ασύλου πλέον, ένα κοινό όραμα. Εάν χάσουμε αυτή την αντιμετώπιση, την αποκοινού, δύσκολα θα καταφέρει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που δεν είναι κατεπήγον απλώς. Είναι φαινόμενο αυτής της ιστορικής περίοδου. Είναι πολύ ε, απλουστευτικό να βλέπουμε το θέμα της μετανάστευσης υπό την οπτική γωνία του κατεπήγοντος, της κατεπήγουσας ανάγκης. Αυτή τη στιγμή διωγμή σε κάποιες χώρες σε αυτό το τεταρτημόριο της υδρογείου από την άλλη όχθη της Μεσογείου η πόλεμη, η αστάθεια της Λιβύης όλα αυτά κάνουν, οδηγούν στην πρόβλεψη και δεν είναι καμιά φοβερή πρόβλεψη ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις θα βρίσκονται δίπλα μας για πάρα πολύ ακόμα, όπως έχει γίνει και σε άλλες ιστορικές περιόδους. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις των 100 μελών και το Συμβουλίο πρέπει να εργαστούν από κοινού, για να υπάρξει μια κοινή θεώρηση. Ως προς την κοινή αυτή θεώρηση να ε, μιλήσω και για το Χαρτούμ. Πιστεύουμε ότι είναι επιτυχία αυτές της προεδρίες, διότι για πρώτη φορά καταφέραμε να ε, έχουμε σε υπουργικό επίπεδο δέσμευση κάποιων χωρών της Ανατολικής Αφρικής και του κέρατος της Αφρικής να δεσμευτούν να συζητήσουν και να μιλήσουν για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων της ε, καταπολέμησης του, της διακίνησης και των μελλοντικών δράσεων όχι μόνο για τον έλεγχο των συνόρων. Εδώ χρειάζεται σφαιρική αντιμετώπιση. Να τονίσω δύο στοιχεία. Πρώτον, κάθε περίπτωση συνεργασίας στα πλαίσια της διαδικασίας του Χαρτούμ ε, προβλέπει την εθελοντική συμμετοχή. Και δεύτερον, κάθε περίπτωση συνεργασίας προβλέπει και τη συμμετοχή των πολυμερών ε, διεθνών οργανισμών ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια βάση θεμελιώδης επί της οποίας θα οικοδομηθεί όλο το υπόλοιπο εγχείρημα. Όμως η βάση είναι αυτή. Σύνορα ε, σημαίνουν και Frontex. Οπότε εδώ εντάσσονται και όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα δώσω μια γενική απάντηση, διότι ήταν επανειλημμένε οι ερωτήσει που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Εγώ προσωπικώς πήγα σε ένα κρύο υπόστεγο του αεροδρομίου της Λαμπεντούζα και είδα τα, ε, τις ορούς νεκρών σε κάτι τσουβάλια και σε ένα από αυτά τα τσουβάλια είδα και μία μάνα με το μωρό της μέσα στο ίδιο αυτό τσουβάλι. Έχουμε αναλάβει από κοινού την ευθύνη δράσης, χωρίς να περιμένουμε παρεμβάσεις από άλλους. Προφανώς, στην περίπτωση αυτή, εννοώ την Ιταλία. Μιλάμε για μια δράση που κόστισε 9 εκατομμύρια το μήνα, διήρκησε τουλάχιστον 12 μήνες και ε, κόστισε συνολικά 114 εκατομμύρια έχουμε ε, διασώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, αλλά δεν μπορέσαμε να τους σώσουμε και όλους. Όχι, διότι βάσει των υπολογισμών μας 499 είναι τα πτώματα που περισυνελέγησαν και πάνω από 500 είναι σύμφωνα με τον όσο λένε οι διασωθέντες τόσοι είναι αυτοί που χάθηκαν στη θάλασσα. Είναι προφανές ότι η αριθμή αυτή δεν είναι ακριβής διότι ε, βασιστήκαμε στην, ε, ε, στις αφηγήσεις των επιβιωσάντων. Ε, ελπίζαμε στο Μάρε Νόστρομ να έχουμε να σώσει όλε τι ανθρώπινε ζωέ, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν ανταποκρίνεται αυτό στην αλήθεια. Το θέμα των σύνορων είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης Διότι δεν ε, υπάρχει στην ιστορία των συνταγμάτων διεθνώς του δικαίου διεθνώς μια ένωση κρατών όπως έχει κάνει η Ευρώπη ως τώρα. Με το Σέγγεν ακύρωσε τα εσωτερικά σύνορα και τελικά έχουν παραμείνει τα εξωτερικά. Το θέμα λοιπόν της Μεσογείου είναι κεντρικής σημασίας και είναι θέμα της ε, το τι γίνεται σήμερα στη Μεσόγειο. Αλλά αν σκεφτούμε το παρελθόν και το μέλλον, θα πρέπει να κοιτάξουμε και να στραφούμε και προ άλλα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η διαρκή μελέτη του θέματο των σύνορων είναι καθοριστική σημασία. Ω προ την διάσωση στη θάλασσα στα πλαίσια των δράσεων τη Frontex. Αυτή η δράση δεν είναι απόφαση τη Frontex. Είναι θέμα της, του ανυπέρβλητου δικαίου τη θάλασσα, πέρα του σεβασμού των ανθρωπίνων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας που θα πει ότι ενώπιον ε, μιας έκκλησης σε βοήθεια μπορεί να κάνει κανείς ότι δεν ακούει. Οι νόμοι της θάλασσας που υπερτερούν οποιοδήποτε νομοθετικό μας αισθήματος και οποιοδήποτε κανόνα τώρα συζητάμε, οι κανόνες του δικαίου της θάλασσας ε, ισχύουν ε, και έχουν συμπεριληφθεί σε όλους τους νομικούς κώδικες. Κανείς δεν μπορεί να τους υπερβεί. Ε, να τους παραβλέψει. Βεβαίως τα σύνορα είναι 30 ναυτικά μίλια, 30 ναυτικά μίλια από τις Ιταλικές ακτές. Όταν υπάρξει έκκληση σε βοήθεια δεν μπορεί κανείς να την παραβλέψει. Είναι προφανές. Σήμερα όμως από όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση Μαρενόστρουμ και ξεκίνησε η περίοδος σταδιακής εξάλληψης με την επαναπροσέγγιση των Ιταλικών σκαφών στα όρια της ακτογραμμής του Σέγγεν και εφόσον όλα αυτά ολοκληρωθούν στο τέλος της χρονιάς, από τότε λοιπόν ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση τρίτων και ε, όταν είχε ολοκληρωθεί η επιχείρηση Ε, η επιχείρηση Μαρενόστρουμ, εκ εκτοτε 3.100 περίπου άτομα διασώθηκαν ε, εφόσον, από τότε που επιστρέψαμε στα 30 ναυτικά μίλια. Κανείς όμως δεν μπορεί να εμπιστεύεται τα λόγια. Όλα αυτά Αυτά είναι κανόνες που έχουν ε, γραφεί επί χάρτου και ε, δεν μπορεί κανείς να παραβεί τις υποχρεώσεις του, κανένας από αυτούς τους οργανισμούς. Ούτε μπορούμε να στεβόμαστε με τις υποχρεώσεις μας. Μίλησα για τις στατηγικές ε, στη συνεργασία με τις Αφρικανικές χώρες, μίλησα για την θάλασσα, ας μιλήσουμε τώρα για την Ευρώπη. Εδώ υπάρχει το θέμα της επανεγκατάστασης, το έθεσαν κάποιοι και είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Είναι ένα θέμα που φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη με τις ευθύνες της και την αλληλεγγύη της. Αυτοί οι δύο πυλώνες ε, πάνε μαζί συμπορεύονται. Ο ένας χωρί τον άλλο και ο άλλος χωρί τον ένα δεν επιτρέπουν να γίνει τίποτα. Η αλληλεγγύη και η κοινή ανάληψη ευθυνών ε, είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό για τον επιπλέον λόγο ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πλέον επονίδιστη, το πιο επονίδιστο ταξιδιωτικό πρακτορείο αυτών αυτής της εποχής ε, τους ε, εμπόρους ανθρώπων που αναγκάζουν όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη να πληρώσουν το εισιτήριό τους. Αυτή την κίνηση πρέπει να εμποδίσουμε ε, προβαλαβαίνοντας οι δολοφόνοι, αυτοί οι έμποροι να μην συνεχίσουν το μακάβριο εμπόριό τους. Στην Αφρική μπορεί να γίνει η πρώτη φάση ε, αλλά θα είναι το πρώτο μισό. Το υπόλοιπο Ευρώπη αναλάβει κοινώς θα γίνει μόνο εφόσον η Ευρώπη αναλάβει κοινώ τι ευθύνε τη. Είναι αυτό λοιπόν μια πρόκληση που μαζί το Κοινοβούλιο, αρχικη κρατών και κυβερνήσεων, επιμέρου κυβερνήσει δηλαδή, το Συμβούλιο, όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί οφείλουν να αναλάβουν σε αυτό το ε, μάτς το, την μπάλα βεβαίως θα την ε, πάρει πρώτα απ' όλα το κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρώπη εφόσον υπάρξει. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα ευαίσθητο ε, με ιδιαίτερη σημασία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ανέφερε και η κυρία Κινίτσι. Η Ιταλική Προεδρία ξεκίνησε την εξέταση τη πρόταση τροποποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό του Δουβλίνου που προβλέπει του κανόνε για την προστασία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ενηλίκων. Είδα, ανηλίκων. Συγγνώμη, είδαμε και το τι προδιαγραφέ προβλέπει η απόφαση του ΔΕΚ την υπόθεση 648 κάθετος 11 για την ε, προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, αλλά και το τι προτείνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαστε σε επαφή και με την εισηγήτρια Βίξτρον για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ένα καλύτερο ε, μια καλύτερη προετοιμασία για την όλη συζήτηση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θέλει να ξεκινήσει όσο δυνατόν ε, συντομότερα ο γύρο τριμερών διαλόγων με το Κοινοβούλιο και προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία για την προστασία των ε, αλλοδαπών ασυνόδευτων ε, ανηλίκων σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση που έθεσε ο πρόεδρος για το Μητρό Επιβατών, το ΔΕΚ και το Συμβούλιο, ιδίω το πιο πρόσφατο Συμβούλιο, σημείωσε ότι αναμένεται τοποθέτηση, λήψη απόφασης και ότι δεν μπορεί να φανεί αδιάλακτο στην τοποθέτησή του. Επαναλήφθηκε η διάθεση συνεργασίας με το Ευρωκοινοβούλιο για να ορίσουμε, να εξεύρουμε μια συμβιβαστική λύση που προσέχτε, προσέχτε με, είναι μια συμβιβαστική λύση για αυτήν την ιστορική χρονική στιγμή. ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας κυκλοφορίας, ιδιωτικού βίου και ασφάλειας. Πρόκειται για τις αρχές που διακυβεύονται, που η κάθε μια έχει τη δική της αυθύπαρκτη αξία και η κάθε μια πρέπει να διαφυλαχθεί, είναι διαφυλαχτέα. Ε, διαφυλαχτέα. Οι κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις που να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Πρέπει να συμφιλιώσουν μεταξύ τους αρχές και αξίες που ε, πρέπει να αποτελέσουν ένα αρμονικό σύνολο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Λιβύης που έθεσε και ο κύριος Φοντάνα. Συμφωνώ, η Λιβύη πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα. Ε, η Λιβύη επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει προσέγγιση υπουργών εσωτερικών αν δεν υπάρξει και μια σφαιρική στρατηγική που να συνδυάζεται με την, πολιτική, με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιου που ε, αναγνώρισε το έργο της Ιταλικής Προεδρίας ως προς το Σέγγεν να πω ότι το έγγραφο που εγκρίνει το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι είμαστε σε μια προηγούμενη σε μια πρώτη φάση και ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις, ε, την πείρα του παρελθόντος για να γίνει το Σέγγεν αποτελεσματικότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε να ε, παραμελήσουμε, μόνο, να παραμελήσουμε και τις κοντινές περιοχές του Σέγγεν και να κοιτάζουμε μόνο τις επιτυχίες μας. Μου τέθηκαν πολλές ερωτήσεις και για τα θέματα της νόμιμης μετανάστευσης. Η κυρία Ντάλη το έθεσε. Είναι κεντρική σημασία. Διότι ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των, λαθ, ροών της μεταναστευσης, της παράνομης μετανάστευσης, με τα όσα κάνουν οι έμποροι, οι διακινητές ανθρώπων, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις νόμιμες μεταναστευτικές ροές. Το κάναμε στο Ιταλικό εξάμεινο με αποφάσεις και συζητήσεις, αλλά κατά την άποψή μας αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να την αναλάβει η Λετωνική Προεδρία. Το έχει ήδη προαναγγείλει στις ε, προθέσεις της για την αλλαγή σκητάλης στο τελευταίο Συμβούλιο. Νομίζω ότι απήντησα σε όλες τις ερωτήσεις και ότι εξήγησα το δεκάλεπτο. Ζητώ συγγνώμη εάν κάποια μικρολεπτομέρεια κάποια ερώτηση δεν καλύφθηκε, αλλά βάσει των σημειώσεων μου νομίζω ότι απήντησα σε όλα. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Πρόεδρε, αν κάτι λείπει από τι ερωτήσεις, ευχαρίστως να σας απαντήσω και γραπτός. Thank you Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ λυπάμαι που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει περισσότερο χρόνο από όσον διαθέτουμε. Ήταν ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εκείνο της Ιταλικής Προεδρίας και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και μας το παρουσιάσατε, και κάνατε τον απολογισμό σας. Η Προεδρία τώρα θα περάσει στα χέρια της Λετωνίας από την 1η Πρώτου 2015 και αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας για το 2014. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη Γραμματεία για τη δουλειά της. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς και τα, όλα τα μέλη, τους ευρωβουλευτές, το προσωπικό, τους βοηθούς. Καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι και ε, μια ξεκούραστη περίοδο διακοπών.